Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσίαση. Εγώ θα αντικαταστήσω τον πρόεδρο Σεϊκεύσκη, ο οποίος θα επανέλθει σήμερα το απόγευμα. Σας προτείνω να ξεκινήσουμε την αρκετά πυκνή αυτή συνάντηση με την ημερήσια διάταξη. Με μια μικρή τροποποίηση στη σειρά των εκθέσεων. Μετά από αίτημα του κυρίου Γιάρ και αφού συμφώνησε και ο κύριος Ρεμπέγκα θα αντιστρέψουμε το 4 με το 5. Γιατί ο κύριος Γιάρ θα πρέπει να φύγει αρκετά γρήγορα και θα ξεκινήσουμε με το 5 για την απαλλαγή δηλαδή για τον Γενικό Προϋπολογισμό 2013. Και μετά θα επανέλθουμε στην κανονική ημερήσια διάταξη, στο σημείο 4 δηλαδή. Ναι, δεν έχετε παρατηρήσεις να κάνετε γύρω από την ημερήσια διάταξη και την αντιστροφή των δύο σημείων 4 και 5 γίνεται δεκτή η ημερήσια διάταξη, συνεπώς και περνάμε στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 22ης Σεπτεμβρίου, 23ης Σεπτεμβρίου και Δευτέρας Οκτωβρίου. Εφόσον δεν έχετε παρατηρήσεις, σας προτείνω να τις έχουμε κάνει δεκτές μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Λοιπόν, γίνονται δεκτά εμπασπέτω. Στα πρακτικά δεν υπάρχουν αντιρρήσει για το σημείο 3, ανακοινώσει του Προέδρου. Να σα πω ότι η συνεδρίασή μα μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Δυνατότητες διερμηνία υπάρχουν για όλες τις προβλεπόμενες γλώσσες, δηλαδή δεν υπάρχουν για τα μαλτέζικα, τα σλοβακικά, τα εσθονικά και τα λετονικά. Και τώρα θα περάσουμε στο 5 λοιπόν, το σημείο του Πέτερ Γιάρ για την απαλλαγή 2013 στον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε ότι σε αιτήσια βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να απαλλάξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εισαγωγικά μετά από την εκτέλεση του προϋπολογισμού τον προηγούμενο χρόνο. Φέτος θα πρέπει να απαλλάξουμε την Επιτροπή από την ευθύνη της για τον προϋπολογισμό 13. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο καλείται να εγκρίνει τους λογαριασμούς της Ένωσης και την χρήση των ευρωπαϊκών πιστώσεων για το 2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των διαφορετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών εκφράζει την άποψή του για την εφαρμογή και εκτέλεση του προϋπολογισμού ε, βασισμένος κυρίως σε ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου της αναλύσης των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου και της συστάσεις του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Συχνά είναι ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να ζητήσει και κάποιες βελτιώσεις στην οικονομική διαχείριση. Θα δώσω όμως πρώτα το λόγο στον κύριο Γιάρ και μετά στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη και θα κλείσει τη συζήτηση ο κύριος Γιάρ. Έχετε το λόγο κύριε Γιάρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κάνατε μια πολύ καλή εισαγωγή στο θέμα και νομίζω ότι σωστό και κατάλληλο είναι ως Επιτροπή Γεωργίας να εκφέρουμε τη γνώμη μας για το θέμα αυτό γιατί μιλάμε για την επιρροή στα θέματα απαλλαγής Μιλάμε για άσκηση επιρροής σε ό,τι αφορά τα θέματα του προπολογισμού. Στη συζήτηση με τους συναδέλφους ε, εξετάσαμε 11 προτάσεις. Καταλήξαμε σε 11 προτάσεις οι οποίες θεωρώ προσωπικά τις οποίες θεωρώ ότι θα πρέπει να καταθέσουμε στην αρμόδια επιτροπή, στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού για να ληφθούν υπόψη στο τελικό κείμενο. Να σας παρουσιάσω λοιπόν τα σημεία αυτά που είναι πολύ σημαντικά. Καταρχά, πρώτο σημείο. Διαπιστώνουμε, δυστυχώς δηλαδή διαπιστώνουμε, ότι σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις ε, αυξήθηκαν το 2013. Αυξήθηκαν λοιπόν, ήταν στο 3,62% στο 2012 στο 2,9%. Αυτές οι διαταραχές λοιπόν σε... είναι διοικητικής φύσεως και αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν χαθεί τα χρήματα ή ότι έχουν σπαταληθεί. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει ε, μία βασική διαφορά. Θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ μεγάλων ε, σφαλμάτων ή όπως είναι η κατάχρηση, η απάτη, οι υπερβολικές ε, πληρωμές και από την άλλη μικρών αντικειμενικών σφαλμάτων μιας και αυξήθηκε ο αριθμός και το ποσοστό σφαλμάτων. Είναι χαμηλής ποιότητας η έλεγχη, δεν είναι επαρκή η ποιότητα ε, στεγανοποίησης των συστημάτων. Κατά τρίτον, διαπιστώνουμε ότι 70% των ε, δημοσιονομικών διορθώσεων που έγιναν και διαπιστώθηκαν το 2013 ε, εστιάζονται σε τέσσερις χώρες. Υποθέτουμε λοιπόν ότι χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις σε αυτές τις χώρες. Τέταρτον, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αξιοπιστία των πληροφοριών για τις πληρωμές όπως αναφέρεται συχνά υπονομεύεται από λανθασμένη και μία ακριβή ε, αναφορά. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολλές φορές διορθώση, διόρθωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους ελέγχους των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών. Άρα δεν γίνονται σωστά οι έλεγχοι και οι αναφορές. Δεν έχει νόημα αν δεν είναι σωστά τα στοιχεία, γιατί στην τελική ανάλυση αυτά θα προκύψουν ως Δεν βοηθάει λοιπόν κανένα να μην γίνεται σωστή αναφορά. Πέμπτο. Αναγνωρίζουμε την ε, όλο και μεγαλύτερη αναστολή πληρωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις οδηγεί σε σφάλματα και σε λήψεις. Έκτον. θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι πολλά μικρά προγράμματα, τα οποία όλοι θέλουμε να, να προχωρήσουν, όπως για παράδειγμα γάλα και απορροκυπευτικά προς τα σχολεία, ότι αυτά τα προγράμματα δεν είναι πάντα φιλικά προς το χρήστη. Και σημαίνουν και μεγάλη γραφειοκρατία. Και άρα δεν είναι επαρκής η αποδοχή και υπάρχουν ε, περιφέρειες που δεν τα εφαρμόζουν γιατί είναι πολύ υψηλή γραφειοκρατία. Ξέρουμε λοιπόν ότι η γραφειοκρατία αυτή οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό σφαλμάτων. Άρα, θα πρέπει να απαλλαγούν αυτά τα προγράμματα από την γραφειοκρατία. Έπτον, ε, έβδομον. Τα προγράμματα αυτά θα έπρεπε ίσως να περάσουν στο δεύτερο πυλώνα της κοινή αγροτικής πολιτικής. Όγδοο. Ζητούμε Ευρωπαίοι υπάλληλοι να μπουν στις εθνικές υπηρεσίες πληρωμών και να είναι υπεύθυνε. Εκεί που δίνει δηλαδή πολύ υψηλό το ποσοστό σφαλμάτων. Όπου υπάρχουν προβλήματα να υποστηρίξουμε τις χώρες με Ευρωπαίους υπαλλήλους, προκειμένου δραστικά να μειωθούν τα σφάλματα. Ένατον, να πιστήσουμε την προσοχή στην Πολιετή διάσταση της αγροτικής πολιτικής και της διαχείρισης της αγροτικής πολιτικής. Και αυτή η οδηγία να μην αλλάξει σε ό,τι αφορά την ε, σταθερότητα η οποία οδηγεί σε μείωση διαρκή των σφαλμάτων. Δέκατο στοιχείο. Διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό σφαλμάτων το οποίο αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο αναφέρθηκε μάλλον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαφέρει σε πολλές περιπτώσεις σημαντικά από το ποσοστό σφαλμάτων που έχει εντοπίσει το ελεγκτικό συνέδριο. Διευκρινήσεις λοιπόν χρειάζονται. Πώς γίνεται δύο διαφορετικές υπηρεσίες να ελέγχουν το ίδιο πράγμα με τις ίδιες αρχές δεν θα έπρεπε να καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Πώς γίνεται να έχει διαφορετικό ποσοστό σφαλμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτό στο οποίο καταλήγει το ελεγκτικό συνέδριο. Πού είναι λοιπόν η αλήθεια. Στη μέση. Θα ήθελα να μας κάνει μια δήλωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας εξηγήσει τα αίτια της διαφοράς αυτής. Εντέκατο στοιχείο. Καλωσορίζουμε τη νέα ρύθμιση για το 2013-2020 σε ό,τι αφορά και τον ορισμό των ε, σχετικών υπηρεσιών πιστοποίησης ε, σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική αναφορά, την καθαρή διόρθωση των δημοσιονομικών και τον ορισμό των σοβαρών σφαλμάτων. Το καλωσορίζουμε και αυτό. Ελπίζουμε να γίνει διάκριση μεταξύ σοβαρών και πιο ήπιων σφαλμάτων. Ε, στο δέκατο ο σημείο Καλώ ορίζουμε την ε, δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον ορισμό και την έννοια του καθαρής διακρατής διόρθωσης, δημοσιονομικής διόρθωσης στον τομέα της γεωργίας σε ό,τι αφορά τη διόρθωση μεμονωμένων πληρωμών. Αυτά λοιπόν ήταν τα 11 σημεία, πολύ γρήγορα και επιγραμματικά και προσβλέπω στη συζήτηση και στα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Merci, <clears throat> monsieur. Σας ευχαριστώ κύριε Γιάννη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε το λόγο. Αλλιώς θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά η κυρία Μαγκίνες έχει ζητήσει το λόγο. Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο έχω ήδη θίξει ε, αφορά στις σχέσεις της Επιτροπής μας με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών σχετικά με τους ελέγχους και την κριτική που ασκείται στην κοινή αγροτική πολιτική. Απαιτείται να έχουμε μια καλύτερη σχέση με τους ε, ε, συναδέλφους μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Ε, υπάρχουν θέματα τα οποία τίθενται μετά από τις αποφάσεις ε, σχετικά με λάθη τα οποία γίνονται στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι ε, επιδοτήσεις κτλ. Πρέπει μάλιστα να σκεφτούμε ότι κατηγορείται μερικές φορές η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών ότι δεν είναι αρκετά αυστηρή Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε καλύτερα μαζί τους, να τους ενημερώσουμε σωστά και αυτό προς όφελος της κοινότητας της γεωργικής ε, και της εξυπηρέτησης των κοινών στόχων. Δεν έχω μια συγκεκριμένη πρόταση να κάνω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι την προσπάθεια να στείλουμε ένα συνεκτικό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αλλιώς θυμάμαι ότι φοβάμαι ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Θα δώσω το λόγο τώρα στην εκπρόσωπο της ε, Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη, την κυρία Μπέιτσον Μίσεν. Euh, Δεν είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω εγώ για την έκθεση ΓΙΑΡ είναι ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 3η Δεκεμβρίου και θα εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό λοιπόν την 3 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ με το 5, τελείωσε το 5, περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο δηλαδή το 4. Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις για την Μολδαβία. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ρέμπεγκα για την τροποποίηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που προτείνουν συγκεκριμένες εμπορικές ρυθμίσεις ε, για την ε, δημοκρατία της Μολδαβίας. Στις 27 Ιουνίου του 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία της Μολδαβίας υπέγραψαν μια συμφωνία σύνδεσης δημιουργώντας μια ζώνη ε, σε βάθος ελευθέρων συναλλαγών ε, που θα διευκολύνει την, ευρωπαϊκή, την οικονομική ολοκλήρωση της Μολδαβίας ε, ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω όμως και του ρωσικού εμπάργου η Μολδαβία έχει προβλήματα στην εξαγωγή ιδιαίτερα σε οπορολαχανικά για, στις αγορές τις οποίες μέχρι τώρα δραστηριοποιείται. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε μονομερώς να απελευθερώσει πλήρως την πρόσβαση στην αγορά για ορισμένα προϊόντα, οποροκυπευτικά, και με αυτόνομο τρόπο λοιπόν έχει διευκολύνει τις ε, εισαγωγές ορισμένων προϊόντων από τη Μολδαβία. Η τροποποίηση η οποία προτείνεται στον συγκεκριμένο κανονισμό δημιουργεί τρία νέα δασμολογικά, τρεις νέες δασμολογικές ενότητες ε, για τα φρέσκα, για τα νοπά ε, μήλα, ε, τα επιτραπέζια στα φύλλα, όπως επίσης και τα φρέσκα δαμάσκηνα, τα νοπά δαμάσκηνα. Είναι μια προσωρινή λύση βέβαια αυτό το σύστημα των αυτόνομων εμπορικών διευκολύνσεων το οποίο θα τερματιστεί αυτόματα στο τέλος του 2015. Είναι μια προσωρινή ενδιάμεση λύση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρέμπεγκα και δεν ξέρω ποια άλλα μέλη θα ήθελαν τον λόγο. Φυσικά θα μπορέσει να πάρει μέρος στη συζήτηση εφόσον το επιθυμεί και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ρεμπέγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η τροποποίηση του κανονισμού που προβλέπει αύξηση των δοσμολογικών ποσοστώσεων μάλλον κατάρτιση των δεσμολογικών ποσοστώσεων για τρει κατηγορίε προϊόντων, νοπά μήλα, Επιτραπέζα σταφύλια και νοπάδα μάσκηνα, λαμβάνει υπόψη τι ανάγκε τη Δημοκρατία τη Μολδαβία στο δύσκολο αυτό οικονομικό πλαίσιο. Γιατί οι αγρότε τη Μολδαβία αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα εξαιτία του ρωσικού εμπάργου. Δεχόμαστε λοιπόν την κατάργηση των δασμολογικών των δασμών για αυτές τις τρει κατηγορίες προϊόντων μετά την επιβολή των ρωσικών κυρώσεων στα ευρωπαϊκά οποροκυπευτικά. Θα σας εξηγήσω για ποιους λόγους αποφάσισα να στηρίξω αυτή την πρόταση τροπολογίας. Θεωρώ καταρχήν ότι η εδαφική ακαιρεότητα είναι πολύ σημαντική και προϋποθέτει μια βιώσιμη και αρμονική ανάπτυξη της, του εδάφους και της χώρας που θα πρέπει να αξιοποιεί τον πλούτο της και το δυναμικό της. Επίσης η εδαφική συνοχή εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Η, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ε, και η σφαιρική και εις συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στις σχέσεις ε, Μολδαβίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, ο δημοσιονομικό αντίκτυπο πρόταση είναι ελάχιστο και οι συνέπειε αυτών των εξαιρέσεων ε, δεν θα επηρεάσουν σχεδόν καθόλου την ευρωπαϊκή οικονομία. Το 2013 ήταν 0,1% οι εισαγωγέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Μολδαβία. Βλέπετε μελιτέα ποσότητα. Ε, οι ποσότητες, επαναλαμβάνω, είναι μικρές. Είναι μικρές ποσότητες ε, σταφυλιών, ε, δαμάσκινων και μήλων που θα εξαχθούν από τη Μολδαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι τελωνιακές αρχές της Ρουμανίας μας ενημέρωσαν ότι έχουμε 32 φορτηγά με σταφύλια, 59 με μήλα και 36 φορτηγά με δαμάσκηνα. Δεδομένου ότι πρόκειται για νοπά φρούτα, δεν πρόκειται να μεταφερθούν σε μεγάλες ποσότητες και άλλωστε οι μολδαβικές αρχές δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν μεταφορά σε μεγάλη απόσταση τέτοιων νοπών προϊόντων. Οπότε τα νοπά αυτά φρούτα κυρίω ε, θα εξυπηρετήσουν γειτονικέ χώρε ε, και δει την Ρουμανία. Γιατί η Μολδαβία δεν μπορεί να διαθέσει ε, τα νοπά τη φρούτα σε απομακρυσμένε αγορέ τη Ιταλία, Σουηδία, εξαιτία του μεγάλου κόστου μεταφορά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα δημιουργηθεί ανταγωνισμός με τους μεγάλους Ευρωπαίους παραγωγούς, γιατί είναι πολύ περιορισμένοι οι πόροι της Μολδαβίας, ακόμη και για τη σήμανση. Τα Ιταλικά μήλα με Ελίντα, για παράδειγμα, έχουν πολύ διαφορετική συσκευασία. Ενώ τα μολδαβικά προϊόντα θα διατεθούν κυρίως σχήμα ε, και κυρίως για τη μεταποίηση, για την παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας και γενικώ μεταποιημένων προϊόντων. Σε ό,τι αφορά την παρούσα κατάσταση τώρα των Ευρωπαίων Γεωργών, η έγκριση της αναθεώρησης του κανονισμού δεν θα επηρεάσει καθόλου τον Ευρωπαϊκό Γεωργικό Κλάδο, γιατί επαναλαμβάνω ε, είναι απειροελάχιστες οι εισαγωγές που θα γίνουν από τη Μολδαβία. Ενώ ο αντίκτυπος πρώτος αυτής για τους Μολδαβούς Γεωργούς θα είναι πολύ θετικός. Επαναλαμβάνω, οι βασικοί αποδέκτες ε, μέχρι στιγμής των προϊόντων αυτών ήταν ε, η Ρώσοι, η Ρωσία και κυρίως ε, γι' αυτό και το ρωσικό εμπάργκο έπληξε ανεπανόρθωτα τους Μολδαβούς Γιώργους. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν είμαι υπέρ της αλλαγής του κανονισμού. Αλλά και η Μολδαβία θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα και αυτό είναι πολύ θετικό γιατί θα γίνουν κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη γεωργία της Μολδαβίας ε, που σταδιακά αναπτύσσεται και σέβεται όλο και περισσότερο τους κοινοτικού κανόνες. Χάρη στην ε, στήριξη αυτή θα βελτιωθούν οι εμπορικές μας σχέσεις με τη Μολδαβία και θα δημιουργηθεί πρόσφορο κλίμα για περαιτέρω εμπορικές ε, συναλλαγές που θα καλύπτουν και άλλα προϊόντα. Και από κοινωνική άποψη η αναθεώρηση του κανονισμού θα έχει πολύ θετικέ κοινωνικέ συνέπειε γιατί θα κρατήσει του γεωργού στην Ήπεθρο εξασφαλίζοντα ε, ένα εισόδημα γεωργικό και για την επόμενη χρονιά. Για μερικές κατηγορίες προϊόντων ε, έχουμε μεγάλη παραγωγή και επειδή η Μολδαβία δεν έχει δυνατότητες αποθεματοποίηση, αποθήκευση αυτών των προϊόντων ε, θα καταστραφούν αν δεν διατεθούν στις γειτονικέ αγορές. Νομίζω ότι με την πρωτοβουλία αυτή δείχνουμε και αλληλεγγύη προ τη χώρα αυτή, λαμβάνοντα υπόψη τι έκτακτε περιστάσει. Ο κύριος Μπομπάκοφ, ο Μολδαβός ε, Υπουργό Γεωργίας, είπε ότι αναγνωρίζει τη δύσκολη κατάσταση και τις έκτακτες περιστάσεις από το ρωσικό εμπάργο. Ευχαριστούμε κύριε Ρεμπέκα για την παρουσίαση της έκθεσης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ντονάνο. Ευχαριστώ. Εστερνίζομαι σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις του εισηγητού για τις ε, μικρές ε, εμπορικές ε, ροές που θα έχει η Μολδαβία, κυρίως με γειτονικές χώρες και δι' τη Ρουμανία. Και δεδομένως έκτακτης κατάστασης συμφωνώ μαζί του. Επειδή όμως ε, εγώ κατάγομαι από μια περιοχή που παράγει μεγάλες ποσότητες μήλων, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια πριν ε, ε, με βάση τις αυτόνομες προτιμησιακές συνέπειες ανοίξουμε την αγορά μας. Διαπιστώσαμε ότι χωρίς έντονες διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη αυξήθηκαν οι δοσμολογικέ ποσοστώσεις με τη Μολδαβία ξεπερνώντα τι αρχικέ συμφωνίε τι συμφωνίε σύνδεση. Περάσαμε από τι 20.000 στου 40.000 τόνου. Και αυτή η αλλαγή τη τελευταία στιγμή έγινε όταν η Ρωσία απειλούσε να επιβάλλει κυρώσει και στη Μολδαβία μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεση που υπέγραψε η χώρα αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις υποχωρήσεις που κάνουμε και τις παραχωρήσεις προς την ε, Μολδαβία, ίσως ε, δημιουργήσουμε στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά κυρίως μήλων, που ούτως ή άλλως είχε πληγεί από τις ρωσικές κυρώσεις, το ρωσικό εμπάργο. Και οι συνέπειες ε, του ρωσικού εμπάργου είναι ακόμη πολύ έντονε και σοβαρέ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των γεωργών. Υπάρχει πρόβλημα συνέπεια μεταξύ τη κοινή γεωργική πολιτική, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη εμπορική τη πολιτική. Δεν είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνουμε τέτοιε ασυνέπειε και συμφωνίε, αλλά θα ήθελα να το επισημάνω και πάλι, ενώ επαναλαμβάνω παραλαμβάνω τη συμφωνία μου με τη θέση του εισηγητού, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή μεταξύ της γεωργικής μας πολιτικής και της εμπορικής μας πολιτικής. Ευχαριστώ κύριε Ντονάνα, κυρία Σάνορα. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο της κυρίας ε, Σάνορα. Disculpa. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για το θέμα αυτό. Καταρχήν, πιστεύω ότι εδώ δεν μιλούμε για τα συμφέροντα των Γιωργών, ούτε των Μολδαβών, ούτε των Ευρωπαίων. Αλλά ψάχνουμε ουσιαστικά φτηνή πρώτη ύλη για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα της μεταποιητικής βιομηχανίας και της αγροεπιστητικής βιομηχανίας και των μεγάλων εξαγωγών και μεγάλων εξαγωγέων. Και όταν λέμε ότι τα προϊόντα αυτά, επειδή είναι νοπά, δεν πρόκειται να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις, με προβληματίζει. Ποιο θέλετε να κοροϊδέψετε με τέτοιους ισχυρισμού. Όλοι γνωρίζουμε ότι Έχουμε σταφύλια, δεχόμαστε σταφύλια από τη Χιλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Χιλή βρίσκεται πολύ πιο μακριά από την Μολδαβία. Ή έχουμε μήλα από την Αργεντινή στην ευρωπαϊκή αγορά, που είναι πολύ πιο απομακρυσμένες χώρες. Όταν λοιπόν υποβάλλετε τέτοια πρόταση, θα πρέπει να τη στοιχειοθετείτε με βάσιμα επιχειρήματα, όχι με ανεδαφικά επιχειρήματα, που είναι ουσιαστικά ένα πρόσχημα, μία δικαιολογία για να δικαιολογήσουμε μία προσπάθεια, μία επιχείρηση που ουσιαστικά εξυπηρετεί τους μεγάλους εξαγωγείς και τις μεγάλες αγοροπιστιστικές βιομηχανίες. Ενώ οι μικρομεσαίες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μολδαβία θα βγουν χαμένοι από την υπογραφή τέτοιων συμφωνιών, όπως συνήθως γίνεται άλλωστε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή δεν είναι καλοδεχούμενη και επί της ουσίας και επί της μορφής. Ο εισηγητής στην ουσία απλά ε, προσπάθησε ε, να δώσει εξηγήσει ανεπαρκής. Είναι μια έκθεση την οποία θα χαρακτήριζα τυφλή ε, επικυρώνει μεν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες δεν έχουν περιεχόμενο. Στην ουσία μας λέει ότι οι τόνοι οι οποίοι θα εξαχθούν χωρίς δασμολογικές επιβαρύνσεις είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι τόνοι των προϊόντων των απορροκυπευτικών. Αυτό είναι σοφιστία γιατί τα προϊόντα αυτά ήδη από το καλοκαίρι έχουν υποστεί στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια σοβαρή μείωση της τιμής τους. Τα δαμάσκηνα και τα μήλα στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης έχουν ήδη απορροφήσει ένα μεγάλο τμήμα ε, του κατεπήγοντος τμήματος των αποζημιώσεων που μπορεί να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, μείωση τιμών, ρωσικού εμπάργο κτλ. Το να καταργεί κανείς τους δασμούς σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι επιδοτεί ο Ευρωπαίος φορολογούμενος την, την γεωργία της Μολδαβίας. Και μάλιστα και με αναδρομικό τρόπο όπως το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ψεύδεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρόταση την οποία κάνει είναι μια πρόταση που ισοδυναμεί μια απάτη αυτοί οι οποίοι έχουν χρηματοδοτήσει τα διαθέσιμα ποσά ε, είναι και οι κάτοχοί τους και η Μολδαβία δεν μπορεί να ωφεληθεί από αυτές τις δυνατότητες. Εκτός αν θέλουμε να βάλουμε τη Μολδαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να το πούμε σε κανέναν. Και ίσως να ξύπνησα σήμερα το πρωί και να είδα ότι η Ευρώπη έχει 29 χώρες. Ο κύριος Μπούντα. Mulțumesc, domnule președinte. Fără doar și poate că susțin... Uh, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ ανεπιφύλακτα με τον εισηγητή μας και θεωρώ ότι ε, είναι πολύ υπεύθυνο και αλληλέγγυο εκ μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το να επέμβει σε αυτή την περιοχή, βοηθώντας τη Μολδαβία. Η γεωργία της έχει πληγεί και ε, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει καταρχήν ε, η χνηλασιμότητα των προϊόντων που εξάγει η Μολδαβία και να μην γίνει μοναδικός αποδέκτης ε, των απολαυτών αυτών φρούτων η Ρουμανία γιατί ήδη η αγορά της ε, υφίσταται μεγάλες πιέσεις και η παραγωγή δαμάσκηνων επίσης έχουν πληγεί από τις ρωσικές κυρώσεις και στη Ρουμανία. Επίσης θα πρέπει να αναλύσουμε διεξοδικά το δημοσιονομικό αντίκτυπο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να επεκτείνουμε τα μέτρα και μετά το 2005. Γιατί μιλήσαμε για σταφύλια που εισάγουμε από τη χιλή. Γιατί λοιπόν να μην εισάγουμε ε, τέτοια φρούτα από μια πολύ κοντινή χώρα όπως είναι η Μολδαβία. Έτσι θα έχουμε και χαμηλότερο κόστος μεταφοράς και χαμηλότερες τιμές των προϊόντων. Πιστεύω ότι θα βρούμε μια λύση πάντως. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη μία θα θέλαμε να βοηθήσουμε τους Μολδαβούς. Από την άλλη όμως τίθενται ορισμένα ερωτηματικά. Ποιος θα πληρώσει τη βοήθεια αυτή. Ποιος θα καλύψει το κόστος αυτής ε, της ρύθμισης. Αυτά θα φύγουν από τον γενικό προϋπολογισμό. Αυτά θα φύγουν από πιστώσεις οι οποίες θα αφαιρεθούν από τον γεωργικό προϋπολογισμό. Ε, ή θα υποστηριχθούν άμεσα οι έμποροι. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν κάποια ερωτηματικά σχετικά με την αλυσίδα της συναλλαγής αυτής και χρειαζόμαστε περισσότερες διευκρινήσεις. Και δεν ξεχνάμε τα προβλήματα που έχουν η παραγωγή των προϊόντων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χαμηλές τιμές με τις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους και τα υψηλά κέρδη των ενδιαμέσων εμπόρων κτλ. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προέρχονται κυρίως από το ρωσικό εμπάργο σε πολλούς τομείς όπως και τον γαλακτοκομικό άλλωστε όχι μόνο στα οποροκυπευτικά. Εν πάση περιπτώσει η πρόταση αυτή είναι θεωρητικά μια χρήσιμη πρόταση ε, σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο διπλωματικό. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε τα τρομερά προβλήματα που αντιμετωπίζουν η παραγωγή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων. Και δεν θα πρέπει να χειροτερεύσουμε την κατάσταση και μάλιστα εις βάρος ενός πολύ συγκεκριμένου μικρού στο μέγεθός του τομέα. Merci σας ευχαριστώ. Είναι καθαρός εξαγωγέας μήλων και η Ρουμανία είναι κατεξοχήν η χώρα που εισάγει τα σλοβενικά μήλα. Ο συγκεκριμένος κανονισμός κατά τη γνώμη μου έχει περισσότερο πολιτική σημασία και προσπαθεί να ενισχύσει, να συσφίξει τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Οι δημοσιονομικές πτυχές ε, είναι ίσονος σημασίας κατά τη γνώμη μου. Η Ρωσία έχει επιβάλει κυρώσεις για τα προϊόντα αυτά στην Ευρώπη, τα απορροκυπευτικά, και οι κυρώσεις αυτές ε, επηρεάζουν τις τιμές ε, των προϊόντων. Και δεν θα χρειαζόταν να υποβάλουμε τέτοια πρόταση αν δεν είχε επιβληθεί το ρωσικό εμπάργκο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει έναν υπολογισμό των ε, ποσοτήτων που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός. Για τι τάξη μεγέθους μιλάμε. Νομίζω ότι θα έχουμε δεκάδες φορτηγά και εκατοντάδες τόνους ίσως ε, προϊόντων, οπών ε, φρούτων που θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Μολδαβία. Πρώτα λοιπόν θέλουμε μία διεξοδική περιγραφή της κατάστασης για να ξέρουμε για τι ποσότητες φρούτων μιλάμε. Αυτό τον υπολογισμό και αυτή την ανάλυση θα πρέπει να μας την κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης κάτι που ανέφερε ο συνάδελφος Μπούντα από την Ρουμανία. Τι γίνεται με την ιχνηλασιμότητα και την ποιότητα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποιότητα γιατί αφορά και την δημόσια υγεία, την υγεία των καταναλωτών. Θα πρέπει να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια που ισχύουν και τους Ευρωπαίους Γιώργους. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση, λέει ο Πρόεδρος, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο ε, χαρακτηρίζεται και από μια γεωπολιτική διάσταση και δεν πρέπει να το αγνοούμε. Αφορά τη σταθερότητα σε μια γειτονική περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια περιοχή που φύγεται από την σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας και μια χώρα η οποία υποφέρει και η ίδια λόγω του προβλήματος της υπερδυστερίας. Συνεπώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη της ε, όχι αυστηρά οικονομικά τυπικά ε, κριτήρια, αλλά να προσπαθήσει να δει το πώς μπορεί να κάνει μία πρόταση ε, με περισσότερα στοιχεία από ό,τι το κάνει μέχρι τώρα. Και λυπάμαι που σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει τις απαντήσεις τις οποίες έχουμε, τις απαντήσεις τις οποίες απαιτούμε, τις ερωτήσεις τις οποίες έχουμε θέσει δεν θα μας τις απαντήσει ουσιαστικά και εφόσον τα μέλη της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής δεν είναι παρόντες, ε, τα στοιχεία ενημέρωσης ε, τα οποία θα έχουμε θα είναι ελλειπή και εκφράζω την ε, λύπη μου γι' αυτό και δεν θα παραλείψουμε να ενημερώσουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής γιατί η κατάσταση αυτή βλάπτει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμεθα είναι ένα περίπλοκο όπως είπα θέμα, είναι ένα πολυσύνθετο θέμα και λόγω ακριβώς της απουσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουσιαστικά θα ξαναδώσω το λόγο στον ε, ε, εισηγητή για να κλείσει την ε, συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. πολλά μπορεί να πει κανείς στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ένα πράγμα είναι αυτό το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Την επιθυμία μας δηλαδή η Μολδαβία κάποια στιγμή να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βρει τη θέση της στο Ευρωπαϊκό Σύνολο. Ταυτόχρονα η δημοκρατία αυτή, η δημοκρατία της Μολδαβίας έχει προχωρήσει σε όλες τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ζητηθεί από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς τον πλήρη σεβασμό ε, των κοινοτικών ρυθμίσεων. Είναι ε, σαφές βέβαια ότι ίσως ε, να μην είμαστε στην καλύτερη χρονικά συγκυρία για την αύξηση των ποσοστώσεων των εισαγωγών από τη χώρα. Και είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προείπαν και οι συνάδελφοι πρέπει να είναι σε θέση να μας ενημερώσει πληρέστερα αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ είμαι στη διάθεση των συναδέλφων και ελπίζω να συνεχίσουμε την πορεία αυτή να έλθουμε πιο κοντά στη Μολδαβία. Συνεπώς να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 7η Νοεμβρίου 12η Μεσημβρινή το επόμενο πλέον σημείο, το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα. Ο κύριος Νίκολσον είναι σε αυτήν τη φάση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος σε μία άλλη έκθεση για την οποία είναι υπεύθυνος. Ως εκ τούτου λοιπόν σας προτείνω να διακόψουμε Ε, για κάποιο χρονικό διάστημα ε, μέχρι τις 10, για 10 λεπτά να διακόψουμε δηλαδή και να συνεχίσουμε μετά με το θέμα του κυρίου Νίκολσον. Ο κύριος Νίκολσον θα είναι εδώ στις 10. Παρακαλώ και εσείς εφόσον το ε, μπορείτε να είστε παρόντες για να συζητήσουμε για τα γαλακτοκομικά. Ο κύριος Φερόν έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Κάποια από τα θέματα είναι στην ημερήσια διάταξη και είναι σε κρεμότητα, ε, γιατί να μην περάσουμε στο επόμενο θέμα. Και υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που έρχονται από πάρα πολύ μακριά και θα πρέπει οι συνεδριάσεις ε, να γίνονται με τον σωστό τρόπο. Σας προτείνω λοιπόν να μην διακόψουμε και να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Κατάλαβα την παρατήρησή σας κύριε Φερό, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι συντονιστές. Ε, δεν είναι για όλους η συνεδρίαση αυτή και προβλέπεται στις 11.30. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να προτείνουμε στην παρούσα φάση κάτι το διαφορετικό. Άλλωστε ο κύριος Νίκολσον είναι και ο ίδιος συντονιστής. και τα υπόλοιπα σημεία θα συζητηθούν το απόγευμα σήμερα. Η κυρία Σένρα. Ευχαριστώ. Έχω να σας υποβάλω μια πρόταση. Θα έλεγα οι επιτροπές που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος, γεωργίας και αλληλείας γιατί να μην συνεννοούνται ώστε να μη συμπίπτουν οι συνεδριάσεις τους. Θα πρέπει κάπως να συντονίσουμε τα χρονοδιαγράμματά μας γιατί αλλιώς θα επαναλαμβάνεται αυτό το φαινόμενο σύμπτωσης ε, των συνεδριάσεων. Σύμφωνα, ευχαριστώ. Νομίζω ότι δίκιο έχετε. Είναι εύστοχο το, το σχόλιο σας. Ε, θα το διαβιβάσουμε και στις άλλες επιτροπές ε, του περιβάλλοντος, της ε, γιατί υπάρχουν ε, θέματα που ενδιαφέρουν και τις τρεις επιτροπές. Και το ζήτημα του προγραμματισμού των συνεδριάσεων ε, δημιουργεί μερικές φορές προβλήματα. Ίσως θα πρέπει να επιληφθεί η διάσκεψη των Προέδρων και να τροποποιήσει κάπως τα ωράρια των συνεδριάσεων για να μην συμπίπτουν οι συνεδριάσεις. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Περιβάλλοντος και Αλλιές συνεδριάζουν την ίδια στιγμή. Καλό θα ήταν να υποβάλουμε λοιπόν αυτό το αίτημα στη διάσκεψη των Προέδρων και να δούμε αν γίνεται να προγραμματίσουμε κάπως διαφορετικά τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, ώστε να μην συμπίπτουν ε, οι συνεδριάσεις, γιατί όλοι μας είμαστε μέλη σε τουλάχιστον δύο επιτροπές. Και πρέπει να τρέχουμε από τη μία στην άλλη. Εδώ το παράδειγμα του κυρίου Νίκολσον που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή μια σημαντική έκθεση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να έρθει εγκαίρος στη δική μας συνεδρίαση. Ας διακόψουμε όμως για λίγα λεπτά. Θα επανέλθουμε στις 10. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση που δείχνετε για αυτή τη σύντομη διακοπή. Merci. Je vous propose de, de reprendre la, la séance. Παρακαλώ, ας συνεχίσουμε. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκολσον που ήρθε στο μεταξύ. Μετά την παρουσίαση που είχε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σας περιμέναμε κύριε Νίκολσον για να συζητήσουμε την έκθεσή σας για το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον απολογισμό της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Γιατί τον Ιούνιο, όπως ξέρετε, του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπει ο οργανισμός ε, της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, υπέβαλε έκθεση για την οργάνωση ε, και την κατάσταση στο γαλακτοκομικό, προϊόν, στο γαλακτοκομικό τομέα με τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Γιατί, όπω ξέρετε, οι γαλακτοκομικέ ποσοστώσει θα εκπνεύσουν τον Απρίλιο του 2015. Θα έλεγα έω και δυστυχώ που θα εκπνεύσουν. Πρέπει λοιπόν τώρα να κάνουμε ένα απολογισμό της κατάστασης του γαλακτοκομικού κλάδου και από οικονομική και από πολιτική άποψη. Για να κρίνουμε κατά πόσο χρειάζονται επιπλέον μέτρα ε, για να αντιμετωπίσουμε την εξάλληψη των ποσοστώσεων. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλία, η οποία συγγετής είναι ο κ. James Nicholson και χωρίς άλλη χρονοτριβή θα του δώσω το λόγο και κατόπιν στους συναδέλφους για να θέσουμε ερωτήσεις στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κόρτ, που είναι ορμόδιο σήμερα για τα θέματα του γαλακτοκομικού τομέα. Κύριε Νίκολσον, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που σας καθυστέρησα όλους, αλλά ήμουν εισηγητής ε, και για τα καινοτόμα τρόφιμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και είχαμε σχετική συζήτηση σήμερα το πρωί. Και το μοναδικό χειρότερο ίσως από το γαλακτοκομικό κλάδο σήμερα είναι τα καινοτόμα προϊόντα. Ο γαλακτοκομικός κλάδος ε, βρίσκεται σε μια πρώιμη φάση σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα και είναι δύσκολο να γίνουν ακριβείς εκτιμήσεις αν ε, εισαχθούν τα μέτρα, αν τα μέτρα που έχουν εισαχθεί ε, είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε κατά πόσο τα μέτρα που έχουν εισαχθεί έχουν εφαρμόσει επαρκώς ή όχι. Και άρα ουσιαστικά βρίσκομαι μεταξύ σκύλας και Χάριβδης. Είναι πολύ απρόβλεπτη κατάσταση για τους επόμενους έξι μήνες και οι αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν σημειώσει πτώση. Έχουμε 0,3% σε ό,τι αφορά τις τιμές σε, τις περσινές. Και αυτή η τάση συνεχίζεται. Συνεχίζουν να πέφτουν λοιπόν τιμές και οι αγορές σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. τα πράγματα μπορεί να φτάσουν ε, έως ε, και 18 έως 20 πένες στον Ηνωμένο Βασίλειο αναλύτρο λίτρο γάλακτος. Το κόστος παραγωγής είναι 25 έως 26 πένες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον όγκο του προβλήματος. Η μείωση λοιπόν σε ό,τι αφορά τις τιμές ε, καθίσταται όλο και πιο προβληματική, μη βιώσιμε και το Κοινοβούλιο στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το θέμα θα πρέπει να επιδείξουμε μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει να αντιδράσουμε με πολύ υπεύθυνο τρόπο. Η παγκόσμια ζήτηση μεν αυξάνεται, αλλά υπάρχει και υπερβολική μεγάλη προσφορά, υπερβολικά μεγάλη προσφορά στην αγορά. σε άλλους κλάδους και οι μεταποιητές ε, πρέπει να πούμε ότι υποφέρουν λόγω της κατάστασης στην αγορά. Στις αρχές του επόμενου έτους λοιπόν ε, βλέπουμε ενόψεις των εξελίξεων στο επόμενο έτος, βλέπουμε ότι ε, πολλά κράτη-μέλη αντιδρούν και πολλά άλλα κράτη είναι κάτω από τις ποσοστώσεις. Και υπάρχουν και οι κυρώσεις ε, που ακόμα πιο πολύ δυσκολεύουν την κατάσταση για το κλάδο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη η χρονική συγκαιρία. Δεν είναι καθόλου δανεική. Θα δημιουργήσει μεγάλη ανασφάλεια στους ε, γαλακτοπαραγωγούς και αυτό που χρειάζεται τώρα ο κλάδος είναι απεγνωσμένα, είναι σταθερότητα. Παρόλα αυτά, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η αντίδραση της αγοράς τον Απρίλιο, τον Μάιο του επόμενου έτους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε αυτά που θα συμβούν τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, υποσχέθηκε στην προηγούμενη κρίση ότι ποτέ ξανά δεν θα έπρεπε, δεν θα αναγκάζονταν ο γαλακτοκομικός κλάδος να περιμένει πάρα πολύ για τέτοια μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν η δέσμευση αυτή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τηρηθεί και να το φροντίσουμε εμείς αυτό. Θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη της ρύθμισης αυτής και να έχουμε χρόνο αντίδρασης. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για να μην δράσουμε. Θα πρέπει να εξετάσουμε ποια μέσα ενδεχομένως να έχουμε στη διάθεσή μας χωρίς να είμαστε ρίζοσπαστικοί στην αλλαγή της πολιτικής και να επαναφεύρουμε τον τροχό. Θα πρέπει να κοιτάξουμε γιατί οι μεταπητές θέλουν επιστροφές εξαγωγών παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκλείσει τη χρήση των μέσων αυτών. Η παρέμβαση είναι πάρα πολύ ε, ήπιο μέτρο και θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση τακτική της ε, κίνησης, της κινητικότητας της αγοράς για να ορίσουμε το χαμηλότερο επίπεδο της αγοράς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Να μας δώσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχετικά στοιχεία και οι αγορές εξαγωγών είναι κλειδί για την επιτυχία της ε, αγοράς. Και κλείνοντας, ε, Πρόεδρε, να πω ότι χρειαζόμαστε ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε του χρόνου, προκειμένου όσοι θέλουν να παράγουν περισσότερο να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, αλλά παράλληλα να προστατεύεται και η αγορά εάν πέσει σημαντικά η τιμή του γάλακτος. Ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστώ κύριε Νίκολσον για την εισαγωγική σας ανάλυση γνωρίζουμε ότι τα θέματα αυτά είναι επίγοντα και ήταν ε, ακριβώς η ώρα να τα συζητήσουμε και στα πλαίσια της έκθεσης πρωτοβουλίας. Εκφράζω την ευχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να συνεισφέρει με θετικό και επικοδομητικό τρόπο στην συζήτηση που πρέπει να γίνουν. Είστε 30 που έχετε ζητήσει το λόγο και γι' αυτό θα ήθελα να σας προτείνω να περιοριστείτε παρακαλώ σε δύο λεπτά. Δύο με δυόμιση λεπτά. Να είστε απλά συγκεκριμένοι εν πάση στα θέματα τα οποία θέλετε να θέσετε για το μέλλον γενικότερα του τομέα. Η κυρία Χέραντς είναι η πρώτη που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις ε, για πολλά χρόνια εξασφάλιζαν ε, αποδεκτό και σταθερό γεωργικό εισόδημα στους κτηνοτρόφους ε, και άξαν τον κόπο και η εξάλληψή τους θα πρέπει να εξεταστεί με νυφαλιότητα και κυρίως να δούμε νέους μηχανισμούς ελέγχου της παραγωγής για να αναχαιτήσουμε την αστάθεια των τιμών και να εξασφαλίσουμε σταθερό εισόδημα στους κτηνοτρόφους. Είναι σημαντικός και ο κοινωνικο-οικονομικός ρόλος αυτών των ε, αυτού του κλάδου, κυρίω σε μειονεκτικέ ή ορεινέ ζώνε. Και παρόλο που είναι το 14% του συνολικού γεωργικού εισοδήματο, φαίνεται ότι δεν το λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνουν τεράστια προσπάθεια εκτινοτρόφοι και έχουν ε, τεράστιε προκλήσει να αντιμετωπίσουν καθημερινά. Και ε, αυτό το ιδηλιακό τοπίο που μας παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της ήδη παρουσιάζει μια πρώτη αδυναμία και μια πρώτη κοιλίδα οι παραγωγοί μερικές φορές ε, αυξάνουν ε, παράλογα την παραγωγή τους ενώ μειώνονται οι εξαγωγές και οι πωλήσει προς ε, τρίτες χώρες όπως η Κίνα και άρα μειώνονται τιμές. Και αν το συνδυάσουμε αυτό με τις ρωσικές κυρώσεις και την κρίση δημιουργεί ένα τοπίο που είναι πολύ μακριά από το ιδηλιακό τοπίο που μας ε, παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε παρατηρητήριο για τις ευρωπαϊκές τιμές. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να προειδοποιούμε έγκαιρα για τις κρίσεις και να εθετούμε τα κατάλληλα μέτρα. Οπότε, για να αξιοποιήσουμε κατάλληλα το παρατηρητήριο θα πρέπει να προσδιορίσουμε ποια είναι τα επίπεδα της κρίσης με βάση δείκτες που θα έχουν θεσπιστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα και επίσης να έχουμε μηχανισμούς πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης γιατί αν οι εκμεταλλεύσεις χάσουν τα περιθώρια κέρδους, ε, δεν θα πρέπει αυτό να το παραμελούν οι δείκτες. Πώς θα εξηγήσουμε στους ε, γαλακτοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους ότι το αποθεματικό της κρίσης το έχουμε εξαντλήσει γιατί μετά τα 86 εκατομμύρια μόνο θα διαθέταμε για την κρίση. Πώς θα εξηγήσουμε στους κτηνοτρόφους ότι τα πρόστιμα για το γάλα θα μεταφερθούν σε άλλα σημεία του προϋπολογισμού, ενώ αυτοί θα πρέπει να πληγούν διπλά, γιατί αφενός την, έχουν αντιμετωπίσει την εξάλληψη των ποσοστώσεων και δεύτερον έχει εξαντληθεί το αποθεματικό της κρίσης, άρα δεν θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σταθερότητα στο γαλακτοκομικό τομέα για να δώσουμε ενάσματα στους κτηνοτρόφους και κυρίως στους νέους να μην εγκαταλείψουν την παραγωγή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σεροσάντος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζουμε, αρχίζει η περίοδος μετά τις 31 Μαρτίου 2015 ε, των νερών, γιατί θα εξελιχθούν οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου οι τιμές γαλακτοκομικών προϊόντων ακολουθούν μια ευθύνουσα πόρια. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, λέει ότι δεν έχουμε μεγάλη μείωση των τιμών παρά τις μειώσεις ε, των εξαγωγών προς την Κίνα. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές μεγαλύτερη ζήτηση ε, στις παγκόσμιες αγορές, αλλά ήδη έχουμε έκτη συνεχή χρονιά που η ζήτηση από την Κίνα έχει μειωθεί και επηρεάζει την αγορά. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι νέες ευκαιρίες της κοινή γεωργικής πολιτικής. Γνωρίζουμε ότι οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις δεν ε, ε, εμπόδισαν τη μείωση των ε, εκμεταλλεύσεων. Έγιναν πολλές προσπάθειες εξυγχρονισμού, αλλά σε μερικές περιπτώσεις, όπως στη δική μου περιοχή στις Αζόρες, είχαμε μείωση των εκμεταλλεύσεων. Θα πρέπει καταρχήν να, να δούμε ποια είναι η αλυσίδα των αξιών. Από την παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση που λαμβάνεται υπόψη, αλλά μας λείπει η διανομή. Και θα πρέπει να αποφύγουμε τη συγκέντρωση για να μην υποχρεώνονται οι παραγωγοί να εκποιούν ουσιαστικά τα προϊόντα του σε πολύ χαμηλέ τιμέ, μερικέ φορέ φορές χαμηλότερες και από τι τιμέ κόστου. Χωρί γαλακτοκομικέ ποσοστό και χωρί έλεγχο τη αγορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα έχουμε αποκέντρωση ή μετεγκατάσταση τη παραγωγή γάλακτο από τι μειονεκτικέ στι πιο ανταγωνιστικέ περιοχέ. Έτσι όμω θα εξουδετερώσουμε όλε τι προσπάθειε οργάνωση. Ε, ε, των ε, γεωργών και κτηνοτρόφων που έγιναν μέχρι τώρα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς ε, και να προσαρμόσουμε και το γαλακτοκομικό τομέα στον ανταγωνισμό των παγκόσμιων αγορών. Επίσης, θα πρέπει να εντοπίσουμε τις πιέσεις που δέχονται οι παραγωγοί. Θα πρέπει να δώσουμε μια συνέχεια στις συστάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και επίσης είναι σημαντικό και θετικό το θέμα της δημιουργίας του παρατηρητηρίου των τιμών, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε προληπτικά, εκ των προτέρων και γι' αυτό θα πρέπει να εξοπλιστούμε με κατάλληλους μηχανισμούς για να προλάβουμε ή να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες ανισορροπίες που χαρακτηρίζουν την αγορά γάλακτος. Ευχαριστώ. Merci, Σας ευχαριστώ. Ένα διαδικαστικό θέμα. Πάνω από 30 ομιλητές έχουν ζητήσει το λόγο. Γι' αυτό σας θέρμο παρακαλώ να μην ξεπεράσετε το δίλεπτο καθένας για να προλάβουν όλοι οι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο. Περιοριστείτε λοιπόν στα ουσιώδη. Παρόλο που το θέμα είναι σημαντικό. Ούκεν το πόλο το έφω. Ο κύριος Κύρτσος. Λέζω, συγγνώμη. Το γάλα έχει κάποια σχέση με το καθεστώς το πολιτικό. Εάν το πρωί σου χτυπήσει την πόρτα ο γαλατάς σημαίνει ότι υπάρχει ένα καθεστώς δημοκρατίας. Εάν σου χτυπήσει την πόρτα αστυνομικό, σημαίνει ότι βρίσκεσαι κάτω από καθεστώς τρομοκρατίας κρατικής. Είναι λοιπόν ένα στοιχείο δημοκρατικότητας στο Γάλα. Πριν από 30 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνιζα ότι εδώ στην Δυτική Ευρώπη έχετε λίμνες από γάλα και βουνά από βούτυρο και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε. Είχα προτείνει τότε να διατεθούν στους φτωχού λαούς αλλά προτιμήσανε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα μετατρέψει σε κουτάκια από γάλα και σε κουτάκια από βούτυρο και να τα μοιράζει στα, στο στρατό, στα σχολεία και στο πρωινό των ξενοδοχείων. Ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Τι θα γίνει με τις λίμνες από γάλα και το, τα βουνά από βούτυρο. Εδώ στην εισήγηση δεν είδα καμία πρόταση συγκεκριμένη για αυτό το λόγο. Υπάρχουν όμως και χώρες με δυσκολία αξιοποίησης του γάλακτος και των προϊόντων παρόλο που έχουν τεράστιες ε, ποικιλίε γάλακτος εκλεκτές όπως είναι η πατρίδα μου τι γίνεται σε αυτή τη χώρα γίνεται το φίρδιν μίγδι η αγελάδα χρησιμοποιείται για όργωση και για μεταφορά με τα κάρα χρησιμοποιείται για κρέας χρησιμοποιείται για γάλα και όλους τους συνδυασμούς αυτούς δηλαδή για 7 με 7 τρόπους επιλέγω με κάτι παρόλο που στην πατρίδα μου υπάρχουν δυο φυλές αγελάδας με παραγωγή μεγάλη γάλακτος και ένας φτωχός βοσκός έμαθε για τις αλπίνες τις πήρε στην πατρίδα μου έφτιαξε μια παραγωγή και τελικά η τράπεζα του τα πήρε όλα και αναγκάστηκε σε αυτο, οδηγήθηκε σε αυτοκτονία γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα εγώ περιμένω από τον εισηγητή να δώσει απάντηση σε αυτό. Merci. Euh, σας ευχαριστούμε κύριε Γλέζο. Μίλησα πριν για το διαδικαστικό, γιατί αν θέλετε να σας κόβω το μικρόφωνο θα πρέπει να περιορίσετε στο δίλεπτο. Ο κύριος Κάστρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σαφές το πρόβλημα εδώ και ο Νίκολσον το παρουσίασε σωστά. Έχουν ε, πέσει οι τιμές, έχουν συντριβεί οι τιμές και από ό,τι φαίνεται η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί σύντομα. Οι αιτίε είναι γνωστές. Έχει υπάρξει μία μείωση της κατανάλωσης που οφείλεται στην οικονομική κρίση. Έχουμε ένα πρόβλημα σχετικά με το ρωσικό εμπάργκο το οποίο έχει οδηγήσει στη μείωση των τιμών των ε, γαλακτοκομικών προϊόντων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε περαιτέρω ε, από αυτά τα οποία τουλάχιστον μας είπε στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο. Νομίζω ότι οι αισιόδοξε προβλέψεις διαψεύστηκαν πλήρως. Εμείς κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ κάναμε κάποιες προτάσεις. Ο Μισελ Ντόντα είχε πει ότι πρέπει να υπάρξει ένας νέος μηχανισμός διαχείρισης της προσφοράς. Δεν έγινε δεκτές οι προτάσεις αυτές, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος του καθεστώτος προστασίας του γαλακτόκτους, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πάρει νέες πρωτοβουλίες και με βάση την προσπάθεια την οποία κάνει ο Τζιμ για δεύτερη φορά ε, θυμίζω ότι ήταν εισηγητής και για το πακέτο για το γάλα, ή ένα πακέτο που δεν έδωσε πάρα πολλές λύσεις στα προβλήματα τα οποία βλέπαμε να δημιουργούνται μετά το τέλος του καθεστώτος των ποσοστώσεων. Πρέπει λοιπόν να ε, ε, κάνουμε μια δική μας πρόταση διαχείρισης της προσφοράς, γιατί με το τέλος ε, του καθεστώτος ε, θα πρέπει να δώσουμε νέα μέσα στους παραγωγούς να διαχειριστούν αυτή την ε, δραματική θα έλεγα διακύμανση εις βάρος τους των τιμών. Σρόιερ μάλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σημαντικά τα καινοτομικά τρόφιμα του κυρίου Νίκολσον. Θα είμαι γρήγορη. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο δράση για τον προπολογισμό. Γιατί είναι κατεπήγον το θέμα και θα πρέπει να ξέρουμε ε, πώ θα αντιδράσουμε, από πού έρχονται τα χρήματα. Και ένα πρωθυπουργό ε, τη Ολλανδία είπε προχθέ ότι, ότι ε, ενδεχομένω να είναι το τέλο αυτό για πολλέ οικογενειακέ επιχειρήσει στην Ευρώπη θα πρέπει να κοιτάξουμε και την Ήπεθρο αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιγόντως ένα σχέδιο δράσης για να δούμε τι θα κάνουμε και με τον προπολογισμό. Merci, Madame Ευχαριστώ, κυρία Μίλλερ έχει το λόγο. Ναι, σήμερα μιλάμε και συζητάμε το πακέτο για το γάλα και τις ε, δυνατότητες που έχουμε να προωθήσουμε τις δέσμες ε, παραγωγών. Στη Γερμανία έχουμε προχωρήσει πολύ καλά. Ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα σήμερα τι γίνεται και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, πώς εφαρμόζονται όλα αυτά οι δέσμες για τους παραγωγούς και τι επιδόσεις σημειώνονται. Στη Γερμανία, κοιτώντας τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες ε, δεσμών ε, παραγωγών, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον μεγάλες διαφορές ε, στις τιμές και παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει δεν υπάρχουν βελτιώσεις ε, σε επίπεδο παραγωγών. Θα πρέπει να κοιτάξουμε όλο τον κλάδο. Λοιπόν, από το γάλα μέχρι το τελικό προϊόν. Και ίσως ε, και τα μη μεταποιημένα προϊόντα θα πρέπει να υποστηριχθούν. Και καθοριστικό στο σημείο θα είναι πώς θα προχωρήσουμε στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί αυτό το πακέτο δεν ε, μου λέει πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις με υψηλής ποιότητας προϊόντων, αλλά οι οποίες δεν μπορούν να συμμετάσχουν επαρκώς στην αγορά. Και μόνο με την συνολική προσέγγιση θεωρώ ότι θα πατήχουμε κάτι σημαντικό. Η επεξεργασία από την αγορά θα πρέπει να είναι και ο στόχος για να υπάρχει συνολική καλλιέργεια και, στις και συνολική παραγωγή και στις μειονεκτούσες περιοχές. Να ληφθεί υπόψη και η σημερινή κατάσταση, αλλά αυτό δεν γίνεται με το τρέχον πακέτο. Ούτε η έκθεση το 2018 θα μας βοηθήσει. Θεωρώ ότι μετά από ένα χρόνο μετά τη λήξη των ποσοστώσεων θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε και το πόσο δραματική είναι η κατάσταση στη Γερμανία είναι σαφές Το κόστος παραγωγής είναι 26,7 ε, λεπτά και αυτή τη στιγμή στη Γερμανία παίρνουν 14 σεντ, 14 λεπτά η παραγωγή και τελικά πωλείται για 29 λεπτά το προϊόν. Είναι δραματική η κατάσταση. Η κυρία Καστινιέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δραματική η κατάσταση και σας ευχαριστώ που τα παρουσιάσατε όλα τόσο επακριβώς. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ αρνητική η κατάσταση. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το soft landing που μας υποσχέθηκε να μας το δώσει. Είναι δραματική η κατάσταση όχι μόνο στις περιοχές ε, εκείνες που είναι πλέον αλλά και στις μειονεκτικές κυρίως, στις ορεινές περιοχές. Και θα υποστούν ακόμα πιο πολλές πιέσεις ως προς τις τιμές. Στην Επιτροπή μας πριν από κάποιο καιρό είχαμε την έκθεση Dorfman για την παραγωγή γαλάκτος στις ορεινέ περιοχές. Την παρουσιάσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ψηφίσαμε την έκθεση. στο κλάδο αυτό δεν έχουμε λάβει τίποτε ακόμη όμως. Δεν έχουμε ούτε μία πρόταση για λύσεις, για το πώ θα επιληθεί η κατάσταση. Ιδιαίτερα στις ορεινέ περιοχές, όπου είναι τόσο σημαντική η παραγωγή γάλακτο, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα παραγωγή για τους εκτροφείς. Το ανέφερε και η κυρία Μούλερ. Οι αλυσίδε παραγωγή κάνουν κατάχρηση και dumping τιμός ξεδιάντροπα. Στην, Αυστρή, στην Αυστρία έχουμε αλυσίδε ευθυνή παραγωγή, ε, μάλλον φθηνό σούπερ μάρκετ, που πουλούν σε εξευτελιστικέ τιμέ το γάλα. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή πλέον, θεωρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει όχι μόνο τον τομέα του γάλακτος, αλλά όλο τον τομέα των τροφίμων και όλο το θέμα του εμπορίου τροφίμων και ε, ενεργά να δράσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Λοαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν χρησιμοποιείτε τον όρο πακέτο γάλα, η δέσμη μέτρο για το γάλα, σταματήστε επιτέλους να χρησιμοποιείτε αυτόν τον όρο. Γιατί Μία συσκευασία ουσιαστικά μας προτείνεται. Ένα μέτρο διάλυσης, εξάλληψης που θα προκαλέσει τη χρεοκοπία των γαλακτοπαραγωγών. Δεν λαμβάνει υπόψη η έκθεση τις εδαφικές επιπτώσεις της πολιτικής σας. Είπατε ότι ε, είναι χαμηλός αντίκτυπος ε, της εξάλληψης των ποσοστώσεων. Τα δύο τρίτα όμως ε, των των κτηνοτρόφων βρίσκονται στις μειονεκτικές περιοχές. Και η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων είναι μικρές ε, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που ακριβώς επιβίωσαν χάρη στις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις. Θα έχουμε απώλεια ενός δισεκατομμυρίου ε, διεξόδων εμπορικών ε, ενώ θα έχουμε μόνο 20 εκατομμύρια αποζημίωση από το ρωσικό εμπάργο, ενώ είμαστε δεύτερη εξαγωγή. Η έκθεση ουσιαστικά ευνοεί τι μεγάλε εκμεταλλεύσει και αποβαίνει βάρο των τοπικών, οικογενειακών, παραδοσιακών ε, μικρών εκμεταλλεύσεων. Σα ερωτώ λοιπόν, μήπω ο στόχο σα ε, είναι να βάλετε λουκέτο στις μικρές ε, εκμεταλλεύσεις γιατί ουσιαστικά παίζετε το παιχνίδι των πολυεθνικών με την πρόταση αυτή. Ο κύριος Κούσμιουκ. Λάθος. Λάθος, συγγνώμη. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ. Το έγγραφο που μας υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έκθεσή της, επικεντρώνεται στην κατάσταση της 13ης ε, Ιουνίου. Είχαμε τότε όμως ε, τέλος της Άνοιξης καλοκαίρι, τα λουλούδια άνθιζαν, η φύση οργίαζε. Τώρα πλησιάζουμε στο χειμώνα και μέσα σε ένα εξάμεινο τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν. Αυτά που ίσχυαν τον Ιούνιο δεν ισχύουν πια. Πολλά έχουν γίνει στην κυνηγεωργική πολιτική. Και Όσα λέγαμε τότε για την εξάλληψη των ποσοστώσεων δεν ισχύουν πια. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, έχει παρούσα κατάσταση στον γαλακτοκομικό κλάδο. Χθες ε, ε, είχα συνάντηση με γαλακτοπαραγωγούς που ζουν σε κοιλάδες, σε ορεινές περιοχές, με ανθρώπους που είχαν επενδύσει πολλά χρήματα περιμένοντας νέες ποσοστώσεις. Σήμερα βρίσκονται σε απόγνωση γιατί δεν ξέρουν πώς θα αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν συνάψει. Και πίστευαν ότι μετά την κατάρριξη των ποσοστώσεων θα μπορούν να παραγάγουν περισσότερο. Αλλά οι κτηνοτρόφοι των μειονεκτικών περιοχών διαρωτώνται πόσο καιρό ακόμη θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου, να χτυπήσει συναγερμό στο γαλακτοκομικό κλάδο. Γιατί αν συνεχίσουμε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, μέσα σε δύο-τρία χρόνια θα εξαλειφθεί πλήρω η γαλακτοκομική παραγωγή στις ορεινέ περιοχές. Και αποκλείεται να προσελκύσουμε νέους στον κλάδο αυτό, γιατί δεν έχει καμία προοπτική. Οι κτηνοτρόφοι δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στην κατάσταση με την ίδια ταχύτητα που έκαναν άλλοι τομεί. Σας απευθύνω λοιπόν έκκληση. Ακούστε τη φωνή των γαλακτοπαραγών τη Ευρώπη που ζητούν πιο ομαλή μεταβατική περίοδο, πιο σαφή έλεγχο της παραγωγής, γιατί αλλιώς ε, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα αρκέσουν για να διασώσουν τους Ευρωπαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Σας ευχαριστώ κυρία Κιλέρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι προλαλήσαντες αναφέρθηκαν στην κατάσταση του γαλακτοκομικού τομέα αν όλοι είχαμε διαβάσει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα διαπιστώναμε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέμε σήμερα. Και είναι πραγματικά περίεργο. Στην έκθεση της, ε, του Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι η κατάσταση του γαλακτοκομικού τομέα στην Ευρώπη είναι ευνοϊκή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές είναι θετικές. Δεν είναι αυτή η γνώμη ούτε του κλάδου ούτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι συμβαίνει. Και πάλι έχουμε ένα κλάδο, το γαλακτοκομικό τομέα, που χάνει το δίκτυο ασφαλείας που είχε με τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις. Τι γίνεται, με αυτή τη δέσμη μέτρων δίνονται κάποια ενάψματα στις οργανώσεις των παραγωγών και στις υποχρεωτικές συμβάσεις που μόνο 12 χώρες ε, τις έχουν εφαρμόσει και μάλιστα 9 μετά τον κανονισμό αυτό. Οπότε, αυτό που προσφέρουμε στο γαλακτοκομικό τομέα είναι κάτι που έχουν ήδη όλοι οι τομείς. Τι λέμε, ε, να σταματήσει αυτή η αστάθεια των τιμών, αλλά αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς. Είχαμε σταθερότητα τιμών εξαιτία των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Όταν θα καταργηθούν, θα επανέλθουμε στην αστάθεια των τιμών, που ούτως ή άλλως μαστίζει όλου του κλάδου. Και η αλυσίδα των τροφίμων, η διατροφική αλυσίδα, ε, θα πληγεί και θα πλήξει ανεπανόρθωτα και τους γαλακτοπαραγωγούς. Χρειαζόμαστε ειδικά νέα μέτρα στη νέα έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα και εγώ να διευκρινιστεί το θέμα των μειονεκτικών περιοχών, γιατί δεν είναι ομοιόμορφα τα χαρακτηριστικά των μειονεκτικών περιοχών. Και αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε σοβαρό αντίκτυπο στις μειονεκτικές περιοχές, χρειαζόμαστε σαφή διαφανή και ομοιόμορφα, ομοιογενή κριτήρια για τις μειονεκτικές περιοχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ριμπέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μία ακόμη φορά μιλάμε για τα μέτρα της δέσμης του πακέτου για το γάλα που είναι εμφανώς ανεπαρκή για το σημαντικό αυτό κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ξεπεράσει την παρούσα αλλά και τη μελλοντική κρίση. Μάλιστα η κρίση οξύθηκε από τις ρωσικές κυρώσεις. Η κατάσταση αυτή έδειξε την ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβλέπει, να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τις ε, κρίσεις. Μόνο κάποια μέτρα τελευταία στιγμή υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρηγορητική αγωγή δηλαδή ουσιαστικά. Τι θα γίνει μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων, ποιο θα είναι το μέλλον του γάλακτος. Ε, με βάση τις ε, οργανώσεις των παραγωγών, η, η τιμή γάλακτος είναι κατά 10 λεπτά χαμηλότερη από τη τιμή παραγωγής, από τη τιμή κόστους. Στις Αζόρες, ε, την πατρίδα μου, που είναι εξόχως απόκεντρη περιοχή, που είναι μακριά από το κέντρο λήψη αποφάσεων, ο γαλακτοκομικό τομέα έχει διαρθρωτικό ρόλο για την οικονομία και έχει οικονομικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ήδη όμως έχουμε βιώσει τις έμεσε ε, επιπτώσεις και του εμπάργου και της ε, μελλοντική ε, εξάλληψη των ποσοστώσεων. Ήδη έχουν πέσει οι τιμές. Και από τον Ιανουάριο έχουν πέσει και οι τιμές και στο κατσικίσιο γάλα. Θα πρέπει κατεπηγόντω να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποτρέψει την εξαιρετική αστάθεια των τιμών και θα γίνει πολύ πιο οξία η κατάσταση μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων. Δεν θα καταφέρουμε να έχουμε μια ισορροπημένη παραγωγή και να αποφύγουμε υπερβολική συγκέντρωση στις πιο παραγωγικές περιοχές. Τα μέτρα της δέσμης ε, για το γάλα είναι πολύ περιορισμένα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το καθεστώ των ποσοστώσεων. Θα πρέπει να συμπληρωθούν αυτά τα μέτρα με νέα μέτρα για να προλάβουμε σοβαρέ κρίσει, να ρυθμίσουμε την εσωτερική αγορά, να, να μπορέσουμε να ελέγξουμε την προέλευση και φυσικά η πρόταση για το παρατηρητήριο γάλακτο και τον τιμό του γάλακτο ε, είναι ανεπαρκής. Σα ευχαριστώ κύριο Ντόρφμαν. Ναι. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση την οποία συζητάμε εδώ, κύριε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαβάζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί ότι είναι καλά η κατάσταση σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τα βλέπουμε όλα μέσα από γυαλιά, μοιοπικά. Γιατί κοιτώντα τι γίνεται στην ε, κατάσταση στην Ευρώπη, στην αγορά και τα προβλήματα που προκαλούνται, ε, αύξηση της παραγωγής ε, Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πόσο προβληματικά τα βλέπει τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν την αύξηση της τιμής παρέμβασης. Νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει ακόμα πιο υψηλή ε, παραγωγή. Θα είναι ακόμα πιο μεγάλα τα κίνητρα. Δεν μας βοηθάει καθόλου λοιπόν στη τελική ανάλυση αυτή η πρακτική. Επειδή κατά το παρελθόν στην προηγούμενη θετία ήμουν εισηγητή για τα θέματα αυτά, όπως είπε και η κυρία Κρόστιγκερ προηγουμένως, νομίζω ότι καλό θα ήταν να ξανακοιτάξουμε το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, κυρίως σε ό,τι αφορά τις μειονεκτικέ περιοχές, τις ορεινές περιοχές. Αναφέρθηκε το θέμα αυτό. Να υποδείξουμε εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ιδιαίτερο στι ορεινέ αυτέ περιοχέ, στι μειονεκτούσε αυτέ περιοχέ θα μπορούσε να υπάρχει ε, μεγαλύτερο πρόβλημα και είναι κατεπήγον να ληφθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα. Εάν θέλουμε να προκληθούν τεράστια προβλήματα στις, για τις μικρές επιχειρήσεις των περιοχών αυτών. Merci. La parole est à Monsieur Beauvais. Ο Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στα συνολικά νούμερα. Το 2014 η αύξηση της γαλακτοκομικής παραγωγής ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι 5%. 5 με 6%. Τι σημαίνει 5 με 7 εκατομμύρια τόνοι περισσότερο γάλα που δεν θα μεταποιηθεί σε τυρί ή άλλα προϊόντα με υψηλή προσθέμενη αξία, αλλά θα γίνει σκόνη γάλακτος, κυρίως για την παγκόσμια αγορά. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Ταυτόχρονα στη Νέα Ζηλανδία θα έχουμε αύξηση κατά 10% της παραγωγής. Οι Ηνωμένε Πολιτείε επίσης θα έχουμε αύξηση παραγωγής 2%. Δηλαδή θα έχουμε στο, στην παγκόσμια αγορά αύξηση από την... Ε, ε, από τις Ηνωμένε Πολιτείες, Νέα Ζηλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση 10 με 17%. Ενώ η ρύθμιση για την αγορά είναι μείον 1 μέχρι 1. Πώς θα απορροφήσει η παγκόσμια αγορά τόσο μεγάλη αύξηση παραγωγής χωρίς μείωση των τιμών. Αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς μείωση των τιμών. Και η ανεύθυνη πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει καταρρύψει και καταστρέψει κάθε μορφή ρύθμισης θα πρέπει να λαγοδοτήσει απέναντι στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους για τη μείωση της uh, τιμής του γάλακτος που θα είναι δραστική την άνοιξη του 2015 είναι ανεύθυνη και η συμπεριφορά των κρατών που αφήνουν την παραγωγή να φύγει. Η Ιρλανδία. Η ε, προβλέπει αύξηση της παραγωγής του γάλακτος κατά 50%. Είναι ένα αλλοπρόσαλο και αλόκοτο σύστημα. Και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ε, που δεν ήταν μέλη της προηγούμενης ε, Επιτροπής Γεωργίας, όταν συζητήσαμε αυτό το θέμα για τις των ποσοστώσεων, είχε υποβληθεί μια πρόταση στα πλαίσια της ενιαίας κοινή οργάνωσης αγοράς από τον κύριο Νταντάν για τον κανονισμό ε, για τις προαιρετικές αποζημιώσεις. Όλοι οι οργανώσεις παραγωγών και, όλες, και όλοι οι συνεταιρισμοί συμφώνησαν με την πρόταση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε το θάρρος ε, να την δεχτεί. Έδειξε ανευθυνότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ουσιαστικά στριμώχνει στον τοίχο τους γαλακτοπαραγωγούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστεί τους γαλακτοπαραγωγούς. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρχεται και να σε υποβάλει μία έκθεση που είναι τελείως ανακριβής και δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην παρούσα κατάσταση. Επίσης, το πακέτο για το γάλα έχει αποδείξει για μία ακόμη φορά ότι είναι άχρηστο και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των γαλακτοπαραγωγών. Οι υποχρεωτικές συμβάσεις δεν εξασφαλίζουν δίκαιες τιμές παραγωγού, ούτε δίνουν διαπραγματευτική ισχύ στους παραγωγούς. Η απελευθέρωση έχει ολέθριες συνέπειες, καταστρέφει μονάδες γαλακτοπαραγωγής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γυρίσει λίγο πίσω και να θεσπίσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη ρύθμιση της παραγωγής και της αγοράς γάλακτος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Merci, Madame Ευχαριστώ, η κυρία Νόικλ. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι πιστεύω ότι καίγεται η αγορά του γάλακτος και είναι σημαντικό να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν δεν μπορούν να παριστάνε ότι το ξέρει. Το ξέρει και θα πρέπει να το ξέρει. Και θα πρέπει να το διαβάζει και στις εφημερίδες. Από τις εφημερίδες ε, μπορούμε να δούμε τι γίνεται στην αγορά του γάλακτος σήμερα. Εμείς τι ζούμε στη Γερμανία και τι θα δούμε και πιο πολύ στο μέλλον. Κανιβαλισμός μεταξύ επιχειρήσεων. Μία επιχείρηση που θέλει να βγάλει το μάτι της διπλανής για να επιπλέψει. Το θέμα είναι ποιος θα σταματήσει πότε. Κάποιες επιχειρήσεις θεωρούν ότι άμα σταματήσει ο γειτονά του, θα ανέβουν οι πωλήσει τους. Και έτσι υπάρχει μεγάλη αίσθηση της αρέσκειας και ακούμε συχνά να κατηγορούν οι μεν τους δε. Αυτή λοιπόν η δυσαρέσκεια θα πρέπει να την ελέγξουμε με κάποιο τρόπο. Για τους συναδέλφους που μίλησαν για τις μειονεκτούσες περιοχές να πω ότι μερικά πράγματα δεν συμφωνώ. Δεν είναι μόνο θέμα των μειονεκτούσεων περιοχών. Είναι ένα πρόβλημα της συνολικής ε, αλυσίδας παραγωγής, της συνολικής ομάδας παραγωγής, που σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο καλείται να παραγωγεί σε τιμές χαμηλότερες και να πωλήσει τιμές χαμηλότερες της παραγωγής. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να συνεχιστεί αυτό. Γιατί οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα είναι βιώσιμες για να μεταφερθούν στην επόμενη γενναία. Θα πρέπει να το σημειώσει αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιτέλους να δράσει, να ενεργήσει. Ευχαριστώ κύριος Ρόισλινγκ. Κύριος sind... Ναι, χαίρομαι γιατί Ακούω στη συζήτηση κάποιοι συνάδελφοι λέγαν ότι άμα καταργηθούν οι ποσοστώσεις θα είναι πιο οικονομική η παραγωγή, θα γίνουν πιο πολλές εξαγωγές. Δεν ακούω τέτοιε φωνές σήμερα. Με την κατάργηση των ποσοστώσεων θεωρώ ότι κάναμε ένα μοιραίο λάθος. Και όποιος ε, περιμένει στο τέλος της έκθεσης να αποφασίσουμε, μάλλον εγώ περιμένω ότι θα πρέπει να, να λάβουμε τελικά μέτρα για να ε, παρέμβουμε στην αγορά. Είναι δραματική η κατάσταση. Και τελικά, τι θα γίνει. Θα ρυθμίσουμε πάλι τις εξαγωγές. Δεν θα έχουμε επιλύσει όμως το θέμα των ποσοστών ε, του συνολικού όγκου. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. βλέπουμε επιχειρήσεις που έχουν διπλασιάσει το, τον αριθμό των αγελάδων τους από 150 σε 300 στη Γερμανία και περιμέναμε ότι τι, θα λυθεί από μόνη η κατάσταση με των εξαγωγών, η Κίνα δραστηριοποιείται επίσης, το πρόβλημα οξύνεται. Το παρατηρητήριο της αγοράς. Έχουμε προτείνει και ένα μέσο για την παρατήρηση και την επιτήρηση της αγοράς. Γιατί να μην το συζητήσουμε. Ανέφερε και ο συνάδελφος Μποβέ τις προτάσεις Δαντάν σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ. Δεν μας βοηθάει. Ούτε βοηθάμε τους παραγωγούς με το να καθόμαστε και να, καταργιώ, να λέμε τι άσχημη που είναι η μοίρα μας. Όχι, θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τα αναγνωρίζει αυτά θεωρεί ότι όλα θα πάνε καλά. Θεωρώ ότι αυτό τελικά θα πρέπει να το υποβάλει ως πρώτη η Επιτροπή μας. Και αυτό περιμένω από τον James Nicholson. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είμαι νέο μέλος του Κοινοβουλίου και αυτής εδώ της Επιτροπής και δεν γνωρίζω ίσως πολύ καλά τις αιτίες που οδήγησαν στην κατάργηση του συστήματος των ποσοστώσεων. Ακούω όμως επανειλημμένα τις ανησυχίες πολλών γύρω από την κατάργηση αυτή και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί τους. Η περίοδος ε, κατά την οποία συντάχθηκε η συγκεκριμένη πρόταση είναι εντελώς διαφορετική από την σημερινή περίοδο και νομίζω ότι ε, μετά την πλήρη εφαρμογή της απόφασης της κατάργησης η κατάσταση θα χειροτερεύσει. Οπότε ή θα καταργήσουμε την σταδιακή κατάργηση του συστήματος των ποσοστώσεων, γιατί θα οδηγήσει πραγματικά σε χάος, ή εάν πράγματι καταργήσουμε το σύστημα θα πρέπει να πάρουμε τις κατάλληλες αντίστοιχες αποφάσεις να φροντίσουμε σαν παράδειγμα την αλυσίδα των πληρωμών όπως λέγεται, να προσπαθήσουμε Ξέρετε το σύστημα που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τη λεγόμενη μήνυμου μη βασική τιμή. Αν δεν κάνουμε τίποτα γύρω από όλα αυτά, τότε τα πράγματα θα χειροτερεύσουν πολύ περισσότερο. Το ρωσικό εμπάργο ε, οδηγεί σε απόγνωση τους παραγωγούς και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Δεν ξέρουν τι θα γίνει με τα προϊόντα τους όταν καταργηθεί και το σύστημα των ποσοστώσεων. Το να χάσει κανείς τις εξαγωγικές του αγορές ε, μέσα σε μια νύχτα είναι κάτι το οποίο συνέβη και το οποίο οδήγησε στη συντριβή των τιμών ουσιαστικά. Ε, η παραγωγή αυτή τη στιγμή γίνεται με πολύ χαμηλότερο κόστος και τα προϊόντα περιμένουν στις αποθήκες να φτάσουν οι τιμές σε επαρκές επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την κατεύθυνση αυτή. Δεν μπορεί να μην έχουμε έναν αμυντικό μηχανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κλείσει πλέον τον κατάλογο των ομιλητών. Όλοι έχουν ζητήσει έτσι και αλλιώς τον λόγο. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Ντονανό και μετά Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής, ο κύριος Νίκολσον, πολύ κανά έκανε και υπενθύμησε την πτητικότητα σε εισαγωγικά και το απρόβλεπτο της αγοράς. Όταν καταργήθηκαν όμως οι ποσοστώσεις, όταν ελήφθη η απόφαση πριν από πέντε χρόνια, πολλοί από εμά προειδοποιήσαμε για τους κινδύνους ε, της ε, απορρίθμισης. Από τη μία βλέπουμε ότι ε, δεν αυξάνεται πια η κατανάλωση, ιδιαίτερα στην Κίνα, και οι τιμές πέφτουν και όχι μόνο εδώ, αλλά και στη Νέα Ζηλανδία και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό λειτουργεί σαν ψαλίδι και θα οδηγήσει σε ακόμα περαιτέρω μείωση της τιμής του γάλακτος. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατανοήσει την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί και να βρει κάποιες λύσεις, γιατί αυτό ε, θα οδηγήσει και σε προβλήματα και στην εκτροφή των βοηδών. Ε, η αγελάδα είναι υποπροϊόν του γάλακτος θα έλεγε κανείς, δηλαδή όταν οι παραγωγοί δεν παράγουν πλέον γάλα, ε, χρησιμοποιούν τις αγελάδες για την παραγωγή κρέατος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στην αγορά του κρέατος και θα έχουμε ένα διπλό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα στο γάλα και ένα πρόβλημα στο κρέας. Θα πρέπει λοιπόν να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προβλέπει, τι μέτρα έχει πάρει για τον τομέα των κρεάτων και τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς για το γάλα. Μήπως πρέπει όπως πιστεύουν πολλοί συνάδελφοι να τεθούν πάλι σε ισχύ μηχανική ρύθμισης. Σμιθ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Και βρίσκομαι σε μια περίεργη κατάσταση, γιατί είμαι εδώ από το 2007 και θυμάμαι την πρώτη έκθεση Νίκολσον που είχαμε το θέμα αυτό, τι συζητήσεις που κάναμε τη Fisher Ball που συζητήσαμε το ίδιο θέμα. Και μου κάνει εντύπωση που οι συνάδελφοι μας λένε ότι είναι καινούργιο το θέμα αυτό. Όχι, είναι τακτικό θέμα, το οποίο συχνά έχει αντιμετωπίσει η Επιτροπή μας. Ακόμα και όταν ο Τζιμ πρωτοεκλέχθηκε, τότε ήδη ήταν πρόβλημα αυτό, δεν το έχουμε λύσει ακόμα θα πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονό ότι πρόκειται για ένα δομικό πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή γαλακτοπαραγωγή. Και οι παραγωγοί επίση θα πρέπει να αποδεχτούν την ευθύνη του για το θέμα αυτό. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα. Εδώ μιλάμε για το ρωσικό εμπάργκο και σε πέντε χρόνια πάλι κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Είναι ένα δομικό πρόβλημα, διαστατικό πρόβλημα. Το πώ παραγάγουμε γάλα και στην Υπηρώ μα και σε όλο τον κόσμο. Η υπερβολική παραγωγή και κάποια κρατημένα δεν βοηθούν καθόλου την κατάσταση. Είναι λοιπόν δομικό πρόβλημα θεωρούν οι παραγωγοί ότι είναι σε ανταγωνισμό με τους ε, γειτονές τους και όχι σε συνεργασία και δεν είναι σωστή η κατανομή της αγοραστικής δύναμης και θεωρώ ότι υπάρχει κατάχρηση σε κάποια το κομμάτια της ε, αλυσίδας εφοδιασμού και μου άρεσαν τα σχόλια του Επιτρόπου Χόγκαν για να υπάρξουν σωστά μέτρα για την αντιμετώπιση του θέματος αυτούς, αλλά θα ήθελα να σας καλέσω να κοιτάξετε το δεύτερο πυλώνα, όπου υπάρχουν διάφορα μέτρα που ε, ενθαρρύνουν την εθελούσια σχηματισμό ε, ενώσεων παραγωγών προκειμένου να μπορέσουν οι θέσεις τους να βελτιωθούν και οι εκπροσώπηση των θέσεων τους στην αλυσίδα ε, εφοδιασμού γιατί μέχρι να λύσουμε το δομικό πρόβλημα το θέμα αυτό θα συνεχίσει να επανέρχεται και πραγματικά δεν είναι καινούριο. Merci. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιο. Να ετοιμάζεται ο κύριος Δαντάμετα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το πακέτο για το γάλα δεν φαίνεται συνοπτικά να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Ε, εξαρτάται από τους όρους της ε, αγοράς σε κάθε κρατος μέλος και τα κίνητρα για τη δημιουργία ενώσεων παραγωγών δεν έχουν πετύχει. Είτε επειδή ήταν πολύ ευνοϊκές οι ε, συνθήκες και οι ώρα πριν από κάνα χρόνο, είτε επειδή πραγματικά δεν θέλουν να συνεργαστούν. Δεν προαγάγεται λοιπόν η αποδοτικότητα και τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο δεν αποσκοπούν στη βελτίωση της ευρωπαϊκής κατάστασης. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν εξειδίκευση, ε, προστιθέμενη αξία τοπικά, αποτελεσματικότητα με τρόπο που να ταιριάζει στους εκτροφείς του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε στις ενώσεις παραγωγών να γίνουν τόσο μεγάλες ώστε να ανταγωνιστούν τα σούπερ μάρκετ γιατί σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Και τι γίνεται με τις πράσινες αγορές γιατί μας λένε ότι υπάρχουν στις αγορές των μέλλοντος ε, μεγάλη αστάθεια. Η αστάθεια υπάρχει και τώρα. Τι γίνεται με την σκόνη γάλακτος. Γιατί ε, έχει, έχει λειτουργήσει το σύστημα αυτό με τα δημητριακά. Γιατί να μην λειτουργήσει και με το γάλα. Χρειάζεται κάποια κερδοσκοπία, χρειάζεται κάποιο μελλοντική, ένα μελλοντικό όρομα. Και τι γίνεται με το φορτίο που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους γαλακτοπαραγωγούς σε ό,τι αφορά την ταφή των ζώων, την τοξικότητά τους και ανοησίες. Είναι τόσο ακριβή η παραγωγή ενέργειας που πλήττει και αυτούς που τροφοδοτούν τις γαλακτοκομικές μονάδες. Έχω κι άλλα να πω, Πρόεδρε, αλλά επειδή μου βάλατε χρονικό όριο θα σταματήσω εδώ. Merci, la parole à Monsieur Dantin. Σε ευχαριστώ, κύριε Dantin, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα του γάλακτος και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου μας έχει απασχολήσει. Δεν θα πρέπει να έχουμε κοντή μνήμη. Ε, κάναμε και ε, παλαιότερα αρκετές ε, προτάσεις για την οργάνωση της αγοράς. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, ανάλογα με την εθνικότητά τους, δεν υποστήριξαν τις προτάσεις αυτές. Και στο Συμβούλιο κάποιες κυβερνήσεις ήταν αντίθετες με τις προτάσεις που κάναμε. Θα πρέπει λοιπόν κάθε κυβέρνηση, ιδιαίτερα αυτές οι οποίες αρνήθηκαν η κοινή οργάνωση αγοράς να περιλαμβάνει ε, ε, δράσεις σε περίπτωση κρίσης στον γαλακτοκομικό τομέα, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και συνεπώς να πάρουν και τα μέτρα τα οποία χρειάζεται. Ένα από τα άρθρα της ε, κοινή οργάνωσης της αγοράς δίνει την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση κρίσης όπως τώρα να κάνει νέες προτάσεις. Αλλά όπως πριν από δύο-τρία χρόνια στα πλαίσια της συζήτησης για το πακέτο γάλακτος, διαπιστώνει κανείς ότι το εγκεφαλογράμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εντελώς επίπεδο. Τι νέα μέτρα έχουμε στη διάθεσή μας, τίποτα. Τι ομάδες εργασίες ειδικέ έχουμε στη διάθεσή μας, τίποτα και συνεπώς υπάρχει θέμα ευθύνης, υπάρχει θέμα ευθύνης και κάποιων πρωταγωνιστών του τομέα. Ήμασταν εδώ στην διάσκεψη που είχε οργανώσει ο προηγούμενος επίτροπος για το χαλακτοκομικό. Ε, και δεν θα ξεχάσουμε την εκστρατεία των ορισμένων βιομηχάνων και επαγγελματικών οργανώσεων που μας έλεγαν ότι η αγορά είναι αυτοδιαχειριζόμενη και δεν υπάρχει ανάγκη να την διαχειριζόμαστε σαν να ήταν σε κρίση. Αυτοί οι οποίοι τα έλεγαν αυτά χτες, σήμερα πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη και να αναλάβουν τις συνέπειες της κρίσης του τομέα. Στο πακέτο για το γάλα υπήρχε και η πρόταση για τη συμβολεοποίηση, η οποία επέτρεπε ε, να υπάρχουν ανώτατα όρια σε περίοδους κρίσης. Ποιες είναι οι χώρες λοιπόν οι οποίες υπονόμευσαν το σύστημα και το συκοφάντησαν, οι χώρες αυτές να μην κλαίνε σήμερα. Αυτοί οι οποίοι πρέπει να κλαίνε είναι η παραγωγή γάλακτος, οι οποίοι πράγματι τους εγκατέλειψαν όλοι γιατί η αγορά, η βασιλείς της αγοράς στην αναζήτηση των κερδών τους αγνόησαν και τώρα χάνουν και τα κέρδη τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντόντα. Ο κύριος Καπούτο έχει το λόγο. Και εγώ τελευταίος ίσως παίρνω το λόγο. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλά έχουν ήδη υποθεί. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω την βαθιά μου ανησυχία για την ε, ικανότητα που έχει το διακανονιστικό πλαίσιο να ανταποκριθεί στο πτυτικό ε, χαρακτήρα της ε, αγοράς και σε μια κρίση η οποία φαίνεται ότι είναι διαρθρωτικού τύπου και ξεπερνά το πρόβλημα των ποσοστώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ε, έχει ήδη διευκρινιστεί στάθηκε αρκετά αδρανής και δεν ε, ε, αξιολόγησε σωστά το μέγεθος των αρνητικών μέτρων του πακέτου για το γάλα. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι το διακανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί σύντομα να αλλάξει. Τίποτα όμως δεν γίνεται για να αλλάξει ένας τόσο σημαντικός τομέας όπως αυτός του γάλακτος, κάτι το οποίο θα έχει από ό,τι φαίνεται και κοινωνικές συνέπειες. Λοιπόν η έκκληση την οποία απευθύνω ε, μαζί με όλους τους άλλους συναδέλφους είναι να ζητήσω από, τους, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει μέτρα το ταχύτερο δυνατόν γιατί όσο καθυστερούμε τόσο ε, θα έλεγα ευνοούμε την καταστροφή του τομέα. Σας ευχαριστώ η κυρία Κανιέτε. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα τιμών και ένα επαρκές εισόδημα για τους ε, παραγωγούς, ιδιαίτερα σε περίπτωση που έχουμε υπερπαραγωγή ή κρίση. Η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας του κ. Νίκολσον για το πακέτο γάλακτος θα πρέπει να περιλαμβάνει λύσεις, μηχανισμούς και μέτρα για να βοηθήσουμε πραγματικά τους ε, παραγωγούς, ιδιαίτερα όταν έχουν πληγεί ε, τα μάλα μετά από άλλες αποφάσεις και πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα κρίση ε, είτε στο γάλα είτε στα απορροκυπευτικά εξαιτία του ρωσικού εμπάργου δείχνει πόσο επιτεκτική είναι ανάγκη στοχευμένων ε, συμπληρωματικών μέτρων και αποζημιώσεων. Και τα μέτρα διαχείρισης της κρίσης και της αγοράς δεν είναι επαρκή αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα τα παραδοσιακά μέτρα διαχείρισης αγοράς, όπως είναι η ιδιωτική αποθεματοποίηση ή παρεμβάσεις, ε, διαπιστώσαμε ότι δεν ε, εξυπηρετούν το στόχο για τον οποίο είχαν ε, σχεδιαστεί. Η κατάσταση για τους Ευρωπαίους γεωργούς και παραγούς όλο και επιδεινώνεται, ιδιαίτερα για τους Φιλανδούς και τους παραγούς της Βαλτικής. Βρίσκονται στο χείλος της χρεοκοπίας αυτοί οι άνθρωποι. Χθε έστειλα ε, επιστολή στον Επίτροπο Χόγκαν και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τον κύριο Γιούγκερ, καθώς και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ζητώντας την ανέβρεση λύσεων, κατάλληλων λύσεων, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης διόρθωσης της κατάστασης. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα αποφάσισε ε, να αφήσει τα κατά 800 εκατομμύρια τα έσοδα ειδικού σκοπού και να τα κατευθύνει σε άλλες πολιτικές. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει δημοσιονομικά να διαθετηθούν και αυτά τα προβλήματα και να καλυφθούν οι ανάγκες, αλλά όχι από, από το αποθεματικό κρίσης για τη γεωργία. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το αποθεματικό για τις ζημίες που προκλήθηκαν από το ρωσικό εμπάργο. Ευχαριστώ. Κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαπιστώνουμε όλοι ότι το πρόβλημα του γάλακτος είναι πολύ Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιληφθεί ότι οι γαλακτοφόρες αγελάδες δεν μπορούν να... Είναι ζωντανά όντα, δεν μπορούν να, να μπουν σε κουτιά. Γι' αυτό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ανάγκε του κλάδου και να προτείνουμε κατάλληλες λύσεις. Φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει αρκετές προσπάθειες ε, για να αναζητήσει νέες ε, αγορές ε, για να διοχετεύσει τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή, λύση θα πρέπει να βρει και... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει και δημοσιονομικές λύσεις, ώστε οι γαλακτοπαραγωγοί ίσως ε, να στραφούν προ στην παραγωγή κρέατος, ώστε να έχουμε και μικτές εκμεταλλεύσεις ε, γαλακτοπαραγωγής και κρέατοπαραγωγής. Γιατί θα πρέπει να εισάγουμε κρέας από την Αργεντινή, ενώ μπορούμε κάλλιστα να το παράγουμε εμείς ίδιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριος Γιάρ. Äh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και την πρέπει να βοηθήσουμε. Έχουν δίκιο οι προηγούμενοι μελητέ. Παρ' όλα αυτά να είμαστε δίκαιοι στη συζήτηση. Διαπιστώνω ότι όλες οι κρίσεις που αντιμετωπίσαμε στο χαλακτοκομικό κλάδο και δεν ήταν λίγε, ω τώρα, δημιουργήθηκαν παρά τι ποσοστώσεις. Και γιατί? Δύο παρατηρήσει, Γιατί οι ποσοστώσεις ω εργαλείο ρύθμιση του όγκου παραγωγή δεν λειτουργήσαν με τις ποσοστώσεις ουσιαστικά επιτρέπαμε πάντα να παράγουμε περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε. Και έτσι λοιπόν ήταν λαθασμένα τα κίνητρα που δώσαμε με τις ποσοστώσεις. Δεν καταφέραμε να, να μειώσουμε την ποσόστοση ως πολιτική, με πολιτική βούληση. Και γι' αυτό Όποιο πιστεύει ότι με τι ποσοστώσει. γιατί σήμερα υπάρχουν ακόμα ποσοστώσει, μην το ξεχνάτε. Αυτό για να είμαστε δίκαιοι. Γιατί δεν πιστεύω ότι ε, αν φύγουν οι ποσοστώσει θα υπάρξει τάξη αύριο. Δύο παρατηρήσει. Κατά πρώτον, η γαλακτοπαραγωγή θα πρέπει να λάβουν την ευθύνη του. την επιχειρηματική του ευθύνη. Πολύ λυπάμαι Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά όλες οι ιδέες που ακούσαμε τότε και στη δική μου περιοχή με μια τιμή α, με τιμή β, με μια σταθερή τιμή, με μια ε, ευέλικτη τιμή, προτείναμε ένα σωρό πράγματα. Δεν έκαναν τίποτα. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή πώς θα παροτρύνουμε τους γαλακτοπαραγωγούς να χρησιμοποιήσουν, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που έχουν για τη διαχείριση κτλ. Δεύτερη παρατήρηση σε ό,τι αφορά τον πυλώνα. τονίστηκε ότι θα πρέπει να αξιοποιούνται πιο πολλοί πυλώνες στην ε, γαλακτοκομική παραγωγή για να βοηθάμε πιο, πολλού, πιο πολύ τους ε, παραγωγούς. Υπάρχουν τα μέσα αυτά, θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Και τρίτον, το αγαπημένο μου το θέμα, κρατικοποίηση Και να μην μένουν και να διαιωνίζονται τα χρέη στον τομέα τη γαλακτοκομικής παραγωγή. Ευχαριστώ κύριε Ντότ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα από το θέμα αυτό που συζητιέται σήμερα. Όταν το έθεσα αυτό για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο, ειλικρινά ήταν πολύ μεγάλη αντίδραση εδώ στην Επιτροπή. Και έκτοτε βλέπουμε ότι αυξάνονται οι πιέσεις στις τιμές του γάλακτος. Η πιο πολύ παραγωγή είναι ρεαλιστές. Αυτό που δεν μπορούν να δεχτούν είναι η συνεχιζόμενη τάση και πίεση επί συνεχιζόμενης ε, χρονικής περίοδου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μεγάλη η θύελα. Έχουμε και τη Ρωσία, έχουμε την αυξηνόμενη παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο και το θέμα της ζήτησης. Έχουμε ποσοστώσεις λέτε και έχουμε και πρόβλημα. Εγώ πρέπει να σας πω όμως πιστεύω ότι είναι μοιραία η περαιτέρω αστάθεια μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων την άνοιξη. Πρέπει λοιπόν και εμείς να δράσουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει. Χαίρομαι λοιπόν που γίνονται και κατεδίαν συζητήσει. Θα ήθελα να ξέρω πώς αξιολογείται Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην αγορά το 2020, πιστεύετε ότι θα συνεχίσει η αστάθεια μέχρι τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει ενδεχόμενες τιμές παρέμβασης και ναι. Και επιστροφές εξαγωγών ενδεχομένω. Η, Ευρωπαϊ... η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να ηγείται των ευρωπαϊκών συζητήσεων. Και θα έπρεπε τουλάχιστον να προβλέψουμε τι θα γίνει με τη μερική κατάργηση των ποσοστώσεων. Στην Βόρεια Ιρλανδία ο τομέα τη καλακτοπαραγωγή είναι και καινοτομικό. Έχουμε ανοίξει νέες αγορές στην Ιαπωνία. Στη Ρωσία είχαμε ξεκινήσει εξαγωγέ πριν το εμπάργο. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Μποβέ, ενδεχόμενη εισαγωγή γάλακτος στην άνοιξη από τις γειτονικές χώρες που επενδύουν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγής μετά το τερματισμό των ποσοστώσεων μπορεί να έχει μοιραίο αποτέλεσμα για τη δική μας, ε, το δικό μας κλάδο και για τη δική μου περιοχή και θεωρώ ότι αυτό μας ανησυχεί ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το βασικό πρόβλημα για πολλούς γεωργούς και δι της ε, Πολωνίας είναι τα πρόστιμα για την υπέρβαση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Για ακόμη μια φορά απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παγώσουν αυτά τα πρόστιμα, αυτές οι ποινές προς τους ε, γαλακτοπαραγωγούς, γιατί είναι τεράστια ζημία ε, και πλήγμα. Έχουν στο κεφάλι τους ε, τη δαμόκλειο σπάθη της, του ρωσικού εμπάργου. Και η αποζημίωση από το αποθεματικό κρίση είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τις ζημίες που υπέστησαν. Και επιπλέον πρέπει να καταβάλουν τα πρόστιμα και τις ποινές εξαιτίας της υπέρβασης γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, παρόλο που με την υπέρβαση αυτή δεν προκάλεσαν καμία απολύτως ε, ζημία. Γιατί δεν έχει γίνει υπέρβαση του συνολικού ποσού των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ποινέ αυτέ τα πρόστιμα αυτά είναι άχρηστα, δεν εξυπηρετούν τίποτα, απλώ πλήττουν του ε, γεωργού και του απειλούν με εξολόθρευση. Απευθύνω έκκληση λοιπόν να παγώσει η καταβολή αυτών των προστήμων. Η κατάσταση στη Φιλανδία, στι βαλτικέ χώρε αλλά και στην Πολωνία είναι εξαιρετικά δεινή για του γαλακτοπαραγωγού δεν θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε τόσο άδικα ενώ ταυτόχρονα έχουμε το ρωσικό εμπάργο που δυστυχώς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει τις ε, απώλειες που προκάλεσε δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ζερκάμπ. Dank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση στον γαλακτοκομικό κλάδο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν προκύπτει επαρκώ από τα εγγραφά. Στην Ολλανδία, στην παρούσα φάση, στο γαλακτοκομικό κλάδο, ε, το μέλλον και βλέπουμε πώ διαμορφώνεται λοιπόν το μέλλον για τον κλάδο αυτό, αν συνεχιστούν οι τάσει αυτέ. Πολύ εκτροφής προετοιμάζονται για την κατάργηση των ποσοστώσεων και βλέπουμε λοιπόν ε, τεράστια αύξηση του αριθμού των ε, ζωών, των, ε, του όγκου των επιχειρήσεων. Αυξάνεται η παραγωγή γάλακτος. Πέφτουν φυσικά και τιμές παράλληλα. Πρόεδρε, η έκταση των στάβλων στην Ολλανδία αυξάνονται, διπλασιάζονται. Χιλιάδες αγελάδες Λέει ένα συνάδελφο από δίπλα ότι αυτό δεν στέκει, αλλά όχι πραγματικά. Έτσι είναι η κατάσταση. Πρόεδρε. Τα ζώα αυτά τα ξεζουμίζουν κυριολεκτικά. Και αυτό είναι επίσης μια παράπλευρη συνέπεια της όλης κατάστασης. Ξέρουμε ότι η παραγωγή γάλακτος ε, δεν είναι και τόσο καλή για την υγεία όσο υποθέταμε παλιά. Και βλέπουμε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει και τα προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Λέμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις μειονεκτούσες περιοχές. Εγώ θεωρώ ότι αντίθετα θα πρέπει να κάνουμε, αντίθετα θα πρέπει να συμπεριφερθούμε θα πρέπει να είμαστε πιο φιδωλοί σε ό,τι αφορά την υποστήριξη μεγάλων επιχειρήσεων και να υποστηρίξουμε τι μικρέ επιχειρήσει πιο πολύ. Ευχαριστώ κύριε Καρτή. Ευχαριστώ πρόεδρε και να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Νίκολσον. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ κρίσιμη αυτή η έκθεση σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το μέλλον του κλάδου γαλακτοπαραγωγής και σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου έναντι τη έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Τα τελικά σχόλια είναι πολύ εύγλωτα. Αναφέρουν ότι η κατάσταση είναι ευνοϊκή και ότι είναι καλέ οι μεσοπρόθεσμες προπτικές στον κλάδο. Αν και αναμένονται επεισόδια αστάθειας τιμής. Νομίζω ότι αυτά τα λέει όλα. Επεισόδια μεγάλες αστάθειες τιμών. Λες και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο και αυτό ξεπεράσει ο κόσμος. Αλλά στην πραγματικότητα κάθε φορά που υπάρχει τέτοια περίοδος αστάθειας, εκτροφής, η ε, μικρή εκτροφής κυρίω, εγκαταλείπουν την αγορά. Και γι' αυτό το παρτίδι για την παραγωγή γάλακτος, το οποίο έχει εφαρμοστεί, θα πρέπει να έχει δυνατότητα να αποστέλνει έγκυρες προειδοποίησεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν προβλέπονται τέτοιες περίοδοι αστάθειας τιμών. Δεν είμαι πεπισμένο ότι τα μέτρα και οι δικλείδε ασφαλεία επαρκούν για να υποστηρίξουν και να προστατεύσουν τους εκτροφείς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα και ελπίζω η έκθεση Νίκολσον να προτείνει μέτρα για να, γίνουν, να εγγυηθούμε τις ελάχιστες τιμές τουλάχιστον. Και αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υποστηριχθούν και να προστατευτούν κυρίω οι μικροί γαλακτοπαραγωγοί. Και να προστατευτεί και το μοντέλο των ε, συνεταιρισμών το οποίο έχει αποδεχθεί τόσο επιτυχές και που έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ καλά τις ανάγκες του γαλακτοκομικού κλάδου. Merci. ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το λόγο. Να υποστηρίξω τον κύριο Γιάρο ο οποίος λέει ότι ποσοστό της γάλακτος ε, θα μπορούσε να είναι ε, μια λύση για μια λιγότερη ασταθή αγορά. Το 2008 ήταν πάρα πολύ χαμηλή τιμή. το 2013 ήταν πολύ ε, καλό έτος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση αυτό που θεωρώ ότι είναι καλό, να μην υπάρχουν ε, εξαγωγών, επιστροφές εξαγωγών. Θεωρώ ότι αυτό είναι απλά μια παράταση του προβλήματος. Θεωρώ λοιπόν καλύτερη, ότι χρειάζεται καλύτερη νομοθεσία. Πιο πολύ περιθώριο για την επιχειρηματικότητα, Natura 2000, και σίγουρα να μην υπάρχουν ποσοστό της γάλακτος, γιατί αυτό αυξάνει και το κόστος και τις τιμές και αυτό, αυτά τα χρήματα καλύτερα να τα δαπανίσουμε για άλλους σκοπούς. Merci. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κορτεκ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μας ε, μιλήσει που φαντάζομαι έλαβε το μήνυμα από τη, για τη σημασία και τη δυσκολία του θέματος. Είναι πολυσύνθετη η κατάσταση στο γαλακτοκομικό κλάδο. Η πραγματικότητα όμως είναι απλή. Ο κλάδος ε, αντιμετωπίζει τεράστιες δυσχέρειες. Φάνηκε από τη συζήτηση ότι ο προβληματισμός είναι ευρύτερος και αφορά το ίδιο το μοντέλο της ε, κοινοτικής γεωργίας. Η έκθεση πρωτοβουλία του κ. Νίκολσον θα είναι πολύ σημαντική και θεωρούμε ότι υπάρχουν δυσκολίες και επιτακτική ανάγκη για λύση του στο συντομότερο δυνατό. Το θέμα επίγει. Διαρωτόμαστε αν ο νέος Επίτροπος Γεωργίας θεωρεί σε μια κατάσταση που συνεχώς επιδεινώνεται ότι έχουμε επαρκή μέτρα και μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Έχετε 10 λεπτά Κύριε Κόρτα, προσπαθήστε να συμπυκνώσετε τις απαντήσεις σας στη σωρία αυτή των ερωτήσεων που δεχτήκατε και περιοριστείτε στα ουσιώδη. Στο τέλος θα δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Νίκολσον για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής και τον κύριο Νίκολσον για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει η Επιτροπή σας για ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τις τελευταίες ερωτήσεις ε, δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω. Δεν είχα τη δυνατότητα να τα συζητήσω τα θέματα αυτά σε βάθος με τον νέο Επίτροπο. Θα πρέπει να του δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο για ένα θέμα ιδιαίτερα περίπλοκο ξεκινάει μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή και νομίζω ότι σίγουρα και σύντομα θα είναι στη διάθεσή σας ο νέος Επίτροπος. Να πω επίσης ότι προφανώς και εμείς θέλουμε να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά περισσότερο μαζί σας και κυρίως με τον κύριο Νίκολσον τους επόμενους μήνες θα προσπαθήσω στον χρόνο τον οποίο μου αφήσατε να δώσω απαντήσεις σε τέσσερις βασικά τομείς. Νομίζω ότι κάνοντας το αυτό θα μπορέσω να ικανοποιήσω όλους όσους έθεσαν τις ερωτήσεις. Καταρχάς η έκθεση δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, στις 30 Ιουνίου, εδώ και 6 μήνες, 5,5 μήνες αφορούσε την λειτουργία του πακέτου για το γάλα. Η συζήτηση και οι προθέσεις άλλωστε και του κυρίου Νίκολσον έδειξαν ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα τα οποία μπορεί να πει κανείς γύρω από το θέμα το συγκεκριμένο. Αυτά τα οποία άκουσα λοιπόν σήμερα το πρωί είναι μια συζήτηση η οποία ξεπερνά σαφώς τα όρια της συγκεκριμένης έκθεσης η οποία, για να είμαι ειλικρινής, ήταν σχετικά περιορισμένη. Και θυμίζω ότι οι προτάσεις οι αρχικές έγιναν με συμφωνία ε, του δικού σας σώματος, το λεγόμενο soft landing, η ήρεμη προσγείωση και η αδυναμία τελικά, απογοητευτικά τα αποτελέσματα της, ε, του τομέα να ενισχύσει τις θέσεις του και να χρησιμοποιήσει ε, τα μέτρα που είχε στη διάθεσή του για τη σταδιακή απόσυρση του συστήματος των ποσοστώσεων. Σχετικά αποτυχία λοιπόν, σχετική αποτυχία, σίγουρα μπορεί να δώσει κανείς νερό στο άλογο λέει ο μιλητής, αλλά δεν μπορεί να το πιέσει για να, να το πιει το νερό αυτό. Ε, υπήρξαν συγκεκριμένες ερωτήσεις στις οποίες απαντήσεις δεν μπορεί να δοθούν. Δεν μπορώ εγώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο γαλακτοκομικός τομέας θα υπακούσει και προφανώς και δεν είναι η Επιτροπή και εγώ υπεύθυνο και υπόλογος για τη συμπεριφορά των γαλακτοπαραγωγών. Τι συνέβη λοιπόν. Τον μήνα Ιούνιο είδαμε ότι κάποιες θετικές εξελίξεις στις τιμές ε, οδήγησαν πραγματικά σε πάνω από 40 σέντ ε, ε, αύξηση ανά 100 κιλά. Βλέπετε λοιπόν ότι υπήρξαν αλλαγές από τότε λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω της μικρότερης ζήτησης από την Κίνα και άλλων προβλημάτων. Αυτά τα ανέφερε και ο κύριος Μποθέ Συνεπώς λοιπόν όλα αυτά συνέβησαν μετά την κυκλοφορία της έκθεσης και χειροτέρευσαν με το ρωσικό εμπάργο που άλλαξε αρκετά τα προβλήματα και η Επιτροπή συμφωνεί με πολλές από τις ανησυχίες που ακούστηκαν σήμερα το πρωί εδώ για το πώς θα λειτουργήσει ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων και πρέπει να προετοιμαστούμε για κάποιους μήνες δυσκολίας στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να αρνηθώ. Και γι' αυτό ε, πολύ σωστά κάποιος από εσά διάβασε την ε, παράγραφο 4 της έκθεσης. Στην φράση αυτή λέγεται ε, ότι οι αγορές είναι ευνοϊκές, οι ε, μεσοπρόθεσμες πρεοπτικές είναι ε, μάλλον ευνοϊκές και το θέμα που πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα της διακύμανσης των τιμών. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν καλές και δεν το λέμε αυτό σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το λένε επίσης και ε, μελέτες από άλλα όργανα. Έχουμε από τη μία λοιπόν τα συγκυριακά στοιχεία της κίνησης της αγοράς, τα οποία αναφερθήκαμε ήδη και ε, από τα οποία υποφέρουμε από το 2008-2009. Και τώρα έχουμε και το εμπάργο το ρωσικό. Να πούμε για το ρωσικό. Επηρέασε ε, το 3% ή κάτω του 3% της ευρωπαϊκής γαλακτοπαραγωγής. Ε, σίγουρα λοιπόν επηρέασε το ρωσικό εμπάργο αλλά όπως είπα και πριν και άλλοι δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε στις συνέπειες του εμπάργου και να μην το χρησιμοποιούμε σαν άλοθη για να πούμε ότι όλα τα προβλήματα στον γαλακτοκομικό τομέα προκαλούνται από το εμπάργο. Δεν είναι αληθές. Αν δει κανείς τις τιμές Πολλοί αναφερθήκατε, πολλά μέλη του Κοινοβουλίου αναφέρθηκαν στις τιμές. Εγώ δεν θα ήθελα να βασίζομαι σε αυτά τα οποία λένε οι εφημερίδες. Εμείς βασιζόμαστε στα μέτρα και στα στοιχεία που μας δίδουν τα κράτη-μέλη. Και εκεί βλέπει κανείς ότι οι τιμές κατεβαίνουν, αλλά υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές οι βαλτικές χώρες χτυπήθηκαν περισσότερο από όλες και αυτό το είπε η κυρία Καλνιέτε. Η κατάσταση εκεί είναι δραματική. Στην Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία μειώσεις τιμών που φτάνουν στο 20% και που είναι πάρα πολύ κοντά στις τιμές παρέμβασης και μπορεί να υπάρξει παρέμβαση πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ σε άλλες χώρες, στη Γαλλία σαν παράδειγμα, η τιμή ήταν συν 4,4% στη Γερμανία μείον 2%, Ρουμανία συν 1,2%, Φιλανδία 0,8 συν. Η κατάσταση λοιπόν δεν είναι εύκολο για μένα έτσι όπως είναι να πω ότι το σύνολο του γαλακτοκομικού τομέα στην Ευρώπη είναι σε κρίση. Δεν έχω τέτοια στοιχεία εγώ. Εγώ ακούω αυτά που λέτε και δεν κλείνω τα αυτιά μου αλλά νομίζω το ότι έχουμε στη διάθεσή μας πιο περίπλοκες, πιο σύνθετες ε, αναλύσεις και στοιχεία μας δείχνουν ένα διαφορετικό πράγμα. Ο Επίτροπος Τσίολος, ο οποίος αποχώρησε πλέον, είχε αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ιδιαίτερα σχετικά με τη Φιλανδία και τις Βαλτικές και είναι θέματα τα οποία εξετάζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνδέεται βέβαια και με την κατάσταση των προϋπολογισμών στην οποία θα επανέλθω σε λίγο. Η εξαφάνιση των ποσοστώσεων σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποχωρεί πλήρως από τον γαλακτοκομικό τομέα και αφήνει πλήρως εκτεθειμένους τις αγορές τους γαλακτοπαραγωγούς. Όχι βέβαια, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε τις άμεσες πληρωμές και φτάνουμε στα 44 δις. Δεν πηγαίνουν όλα στο γαλακτοκομικό τομέα βέβαια, αλλά στήριξη εισοδήματος υπάρχει, η οποία είχε προβλεφθεί για να αντισταθμίσει τη μείωση της τιμής παρέμβασης. Και είχαμε χρόνια με υψηλές τιμές, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει στήριξη λοιπόν και στα πλαίσια της ανάπτυξης της υπαίθρου, ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές, Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα διαθέσιμα μέτρα τα οποία επιτρέπουν το top-up κατά 2,50 ευρώ ανά εκτάριο περίπου. Εν πάση περιπτώσει και εδώ κάνουμε τις καλές προτάσεις αλλά δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε. Ε, τα κράτη τα ίδια είναι αυτά που θα αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες πιστώσεις στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Έχουμε και το δίκτυο ασφαλείας και απαντώντας σε πολλές ερωτήσεις γύρω από όλα αυτά. Θα ήθελα να πω ότι έχει ξεκινήσει ένα εργοτάξιο για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας προμήθειας των τροφίμων. Πώς μπορούμε εμείς από κοινού σε επίπεδο ένωσης να ενισχύσουμε την θέση του παραγωγού στην αλυσίδα της προμήθειας του τροφίμου. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το ανέφερε και ο κύριος Νίκολσον στην αργή της συζήτησης. Κάτι θα πρέπει να γίνει στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό συνδέεται επίσης και με κάποια άλλα στοιχεία τα οποία συζητήθηκαν στα πλαίσια της κοινή οργάνωσης της αγοράς, επιτρέπουμε εξαιρέσεις από τους κανόνες του ανταγωνισμού, άλλο ένα σημαντικό πεδίο, θα έλεγα, εργασίας, το οποίο ερευνούμε προσεκτικά στο εσωτερικό της Επιτροπής. Στρεβλές εμπορικές πρακτικές είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τη, τους παραγωγούς. Έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ειδικά γι' αυτό. Αλλά δυστυχώς για μια ακόμη φορά οι μεγάλες γαλακτοκομικές οργανώσεις δεν θέλουν να πάρουν μέρος. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να φύγετε από εδώ λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ξανά το λάθος να λέει ότι τα πράγματα είναι όλα ρόδινα. Όχι, προβλήματα υπάρχουν. Σας διαβεβαιώ ότι τα προβλήματα αυτά είναι ε, προτεραιότητα για τον Επίτροπο Χόγκαν. Θα επανέλθουμε σε όλα αυτά. Σημείωσα αυτά που είπατε και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Κόρτε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Νίκολσον. Κύριε Πρόεδρε, είπα στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις ότι ήμουν μεταξύ σκύλας και χάριδες. Τώρα θεωρώ ότι είμαι μεταξύ σφύρας και άκμονος, γιατί μετά από αυτά που ακούσαμε στη σημερινή συζήτηση, ενισχύεται η πεποίθησή μου ότι κάτι πάει πολύ στραβά, κάτι είναι πολύ σαθρό σε ολόκληρο το γαλακτοκομικό τομέα. Ο Όλεν Σμιθ είπε πολύ σωστά ότι το έχουμε ξαναδεί το θέμα. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε. Το ακούσαμε πολλές φορές και στο παρελθόν και οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις δεν έλυσαν ε, κατά ανάγκη όλα τα προβλήματα των γαλακτοπαραγωγών στην Ευρώπη. Θα πρέπει και αυτό να το αναγνωρίσουμε. Με την άρση όμως των ποσοστώσεων με τον τρόπο που έγινε. Γιατί η απόφαση για την εξάλληψη των ποσοστώσεων έγινε το 2005-2006 επί Μαριάν Φίσερ Μπολ. Τότε που ο γαλακτοκομικός τομέας βρισκόταν σε πολύ ευνοϊκή κατάσταση και επικρατούσε γενική εφορία. Μετά όμως είχαμε την κρίση του 2008-2009 και τώρα φαίνεται ότι έχουμε μια νέα κρίση. Γιατί δεν λάβαμε δέοντος υπόψη την προηγούμενη. Και τώρα ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι μπορούμε να πάμε το άλογο στην πηγή, αλλά δεν μπορούμε να το αναγκάσουμε να πιει νερό. Αλλά ίσως το νερό που δίνει στο άλογο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να είναι ακατάλληλο, για αυτό το άλογο δεν θέλει να πιει. Ίσως δεν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλη τη σοφία που απαιτείται και ίσως θα πρέπει να συνεργαστεί πιο στενά με την Επιτροπή μας και να εμπλουτιστεί με τις δικές μας ιδέες στο μέλλον. Και κάτι που με απογοητεύσει την προηγούμενη επιτροπή ήταν ο τρόπος που χειρίστηκε το αποθεματικό κρίση για τη Γεωργία. Ήταν πραγματικά αξιοθρύνητος, απαράδεκτος αυτός ο τρόπος και αποτέλεσμα είναι να είναι το Ταμείο Μείων. Και αν αντιμετωπίσουμε πρόβλημα την Άνοιξη, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα να το λύσουμε. Και έχουμε και την ε, υπερισφορά, το super levy, που δημιούργησε ανησυχή στην Ευρώπη, αλλά δεν έδωσε λύσεις. Και ούτε μου αρέσει αυτή η πρόταση να εισπράξει υπερισφορά και να τη διαθέσει σε άλλους τομείς. Αν θέλετε να εισπράξετε περισφορά, τουλάχιστον να τη διαθέσετε για μέτρα στο γαλακτοκομικό τομέα. Αυτός να αποφεληθεί. Και μιλήσαμε για την απαλή, την ομαλή προσγείωση. Μας το είχε πει και η τότε επίτροπος Μαριάν Φισελμπόλ. Αλλά ακούσαμε την ομαλή προσγείωση, αλλά ακόμη να τη δούμε. Ακόμη την περιμένουμε. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον κλάδο για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να τα βγάλουν πέρα. Δεν ακούσαμε ιδιαίτερα σήμερα το θέμα της ισχύω των ε, μεγάλων αλυσίδων παραγωγής των σούπερ μάρκετ, των πολυεθνικών. Γιατί ε, βλέπουμε ένα δύο λίτρα γάλα να στοιχίζει μια λίρα. Ενώ το νερό είτε με είτε χωρίς ανθρακικό είναι πιο ακριβό, 1,5 λίρα. Πώς είναι δυνατόν το γάλα να είναι φθηνότερο από το νερό. Δεν υπάρχει σύγκριση εδώ πέρα. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε μεγαλύτερο ρεαλισμό στον τρόπο διαμόρφωση των τιμών. Και για τους παραγωγούς στις ορεινές και μειονεκτικές ζώνες δεν είναι ίδιο το πρόβλημα. Ξέρω ότι πολλοί λένε ότι το πρόβλημα θα διαθετηθεί με επαναδιάθεση των κονδυλίων του δεύτερου πυλώνα. Μπορεί κάπως να μετριαστεί, αλλά δεν είναι λύση αυτή, γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο για να κρατήσουμε ζωντανές τις ορεινές και τις μειονεκτικές περιοχές. Και το πρόβλημα μας απασχολούσε και στο προηγούμενο πακέτο για το γάλα και με το σημερινό και φαντάζομαι θα μας απασχολήσει και στο μέλλον θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην μου λέτε τι δεν μπορώ να κάνω. Πείτε μου τι μπορώ να κάνω και ας το κάνουμε επιτέλους από κοινού. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ κύριε Νίκολσον. Δεν καταλήξαμε φυσικά συμπέρασμα. Τώρα ξεκίνησε η συζήτηση επί της έκθεσης πρωτοβουλίας. Θα έχουμε στις 21 Ιανουαρίου ε, τη εξέταση του σχεδίου έκθεσης και όπως είπατε είναι καρπός συλλογικής προσπάθειας. Το διακύβευμα είναι τεράστιο και θα πρέπει να βρούμε το μοντέλο που είναι το κατάλληλο για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Σας ευχαριστούμε κύριε Κόρτε για κάποιες απαντήσεις που δώσατε. Θα ήθελα τώρα να διακόψω τη συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε στις 3 με τον κύριο Σεκέσκη που θα αναλάβει και πάλι την Προεδρία. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Φίσλερ για την ενημέρωση που θα μας κάνει για τη Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου, την Expo 2015. Ενώ σε λίγο στις 12 παρατέταρτο θα ξεκινήσει την ίδια αίθουσα η συνεδρίαση των συντονιστών. Καλό μεσημέρι στους υπόλοιπους